Ένα λεπτό για να ολοκληρώσουμε τα της αναφοράς. Ένα λεπτό, παρακαλώ. Ωραία. Και ζητούμε η Επιτροπή των ε, Αναφορών πρώτα-πρώτα να απευθυνθείτε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξεταστεί το αν τηρούνται ή όχι τέσσερις ε, οδηγίες για το νερό, για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, για τα ε, άγρια πουλιά και για τα υπόγεια ύδατα. Οπότε θέλουμε να γίνει κάποια διερευνητική εξεταστική επιτροπή. Να πάρετε στην Δονιάνα και να δείτε από κοντά το πώς παραβιάζονται αυτές οι τέσσερις οδηγίες. Και να δείτε γιατί όλοι οι κοινωνικοί φορείς και οι επιστημονικοί είμαστε κατά αυτών των έργων. Θα πρέπει να αφουγκραστείτε τους Ευρωπαίους πολίτες. Έχει δώσει τόσους πόρους για την προστασία της Δονιάνα η κοινότητα. Άρα θα πρέπει επίσης κάτι να κάνετε τώρα για να ε, σωθεί αυτή η περιοχή και αυτό είναι προς το συμφέρον όλες τις ε, Ένωση. σά ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρόκειται για κάποια υπόθεση που μα είναι πάρα πολύ οικία. Έχει συζητηθεί δύο φορέ στην Επιτροπή. Θα ήθελα να δώσω το λόγο και στον κύριο Γκονσάλες Πραι, προς, ε, ο αναφέρον της αναφοράς 85. Έχετε το λόγο και εσείς για πέντε λεπτά μέγιστο. Uh, Το συγγνώμη, λέει η πρόεδρος, μήπως δεν έχει έρθει ο αναφέρον της δεύτερης αναφοράς. Όχι. Εντάξει. Δεν ήρθε. Οκ. Επομένως θα ζητήσω από τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ε, εκφράσει τη θέση της σε σχέση με την αναφορά 51, ο κύριος Γκόμες. Muchas gracias, señora Presidente. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Σωστά είπατε. Πρόκειται για μια υπόθεση που τη γνωρίζει καλά η Επιτροπή σας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανειλημμένα έχει εξηγήσει την τοποθέτησή της και επίσης έχουμε δημοσιεύσει σειρά ανακοινώσεων. Και αφορούν αυτέ τι εγγενώσει το τι έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τα όσα έχουν καταγγελθεί. Και όπω ήδη έχουμε εξηγήσει, πρώτα-πρώτα έχουμε την ε, οδηγία για την οδηγία του ε, οικότοπου που δεν ε, προβλέπει τίποτα για αυτέ τι περιοχέ που αφορούν το Natura 2000 παρόλα αυτά όμως υποχρεώνει η οδηγία πριν εγκριθούν αυτά τα σχέδια και προγράμματα οι αρμόδιες αρχές να εξασφαλίσουν το ότι αυτά τα έργα δεν πρόκειται να παραβλάψουν αυτές τις ε, περιοχές. Και αυτό κατόπιν αξιολόγησης των επιπτώσεων του, του κάθε έργου σε σχέση με το Natura 2000. Και όπως σας έχουμε ενημερώσει, αποφασίσαμε να ξεκινήσει έρευνα, ούτως ώστε να εξηγηθεί από πλευρά των Ισπανικών αρχών ό,τι χρειάζεται και ο, κάθε λεπτομέρεια που χρειάζεται για το εάν έχει υπάρξει συμμόρφωση με το κοινωτικό δίκαιο όσον αφορά το περιβάλλον. Αποτέλεσμα της έρευνας ήταν το ότι μας ενημέρωσαν τελικά οι αρχές ότι υπάρχουν εδώ τέσσερα έργα για την εξόριξη, την αποθήκευση, μεταφορά του φυσικού αερίου στην Τονιάνα έχει γίνει αξιολόγηση όλων αυτών των έργων όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Και επισυνάπτεται σε αυτές θετική εκτίμηση ως συμπέρασμα. Έγινε αξιολόγηση των περιοχών του Natura 2000. Το συμπέρασμα είναι ότι πουθενά δεν έχουμε κάποιο είδους σημαντικές επιπτώσεις για το Natura 2000 και τις περιοχές του. Μόνο το έργο Μαρίσμα Οξιδεντάλ εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 16 από αυτά τα τέσσερα έργα. Υπήρχε και εκεί θετική αξιολόγηση επιπτώσεων του Σεπτεμβρίου του 10 και η έγκριση δόθηκε επίσης τον Νοέμβριο του 10. Έχουμε τώρα άλλα τρία σχέδια και προγράμματα που ακόμα δεν έχουν τύχει έγκρισης. Οι δε περιφερειακές αρχές της Ανταλουσίας θεωρούν ότι δεν γίνεται να δοθεί για τα άλλα έργα ε, έγκριση δεν δόθηκε άδεια γι' αυτό όσον αφορά το περιβάλλον γιατί ακριβώς υπάρχουν επιπτώσεις όσον αφορά το περιβάλλον. Δεν έχουμε άλλες πληροφορίες για τα άλλα έργα, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει χορηγηθεί καμία έγκριση. Επίσης, μας είπαν οι Ισπανικές Αρχές ότι η έγκριση του Μαρίσμα οξιδεντάλ, όπως και η απόρριψη της αίτηση για το Μαρίσμα Οριεντάλ, ήταν αντικείμενο προσφυγών διοικητικών και στην πολιτική δικαιοσύνη. Οπότε από δεν προβλέπεται να παρέμβουμε ακριβώς μια που κρίνεται η υπόθεση ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων. Δεν έχει διαπιστωθεί παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας από κοντά παρακολουθούμε τις εξελίξεις να δούμε τι αποφάσεις θα ληφθούν και να, για να δούμε τι τύχη θα έχουν αυτές οι προσφυγές. Θα σας ενημερώσουμε. Πρόεδρος. Has Mr. Gonzalez Ο κύριος Γκονσάλες έχει έρθει. Όχι, ωραία. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στα μέλη της Επιτροπής ξεκινώντας από την ε, Κύριε Αλβιόλ. Πρώτα πρώτα ευχαριστούμε τους αναφέροντες και την πλατφόρμα να σώσουμε την Τονιάνα. Σε ευχαριστούμε για το έργο το οποίο έκαναν για την προστασία αυτού του εθνικού πάρκου. Τονίστηκαν δύο πολύ σημαντικά σημεία. Πρώτα-πρώτα ότι δεν έχουμε τώρα κάποιο είδους έργο κοινού γενικού συμφέροντος, αλλά πρόκειται για κίνηση κερδοσκοπική ε, εταιρεία που απλώς θέλει να κάνει δουλειές. Αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη γιατί κινούμεθα σε αυτό το πλαίσιο. Επίσης, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε παράβαση της ε, κοινοτικής νομοθεσίας για και έχουμε αυτά τα τέσσερα έργα. Έγιναν χωριστά οι μελέτες επιπτώσεων. Δεν ελήφθη υπόψη το σωρευτικό αποτέλεσμα και των τεσσάρων μαζί. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη σχετική οδηγία και επίσης είπαμε ότι έτσι είναι δυνατόν τα ύδατα να μολυνθούν και να ρηπανθούν. Και ισχύει σχετική οδηγία. Μιλούμε για εθνικό πάρκο, είναι γενικότερου ενδιαφέροντος. Έχουμε το δίκτυο επίσης ε, το και έχουμε επίσης την οδηγία για τα, εκτός από τα ύδατα την οδηγία για τα πουλιά και επίσης έχουμε την σεισμολογική μελέτη του Πανεπιστημίου που λέει ότι εκεί πέρα υπάρχουν και εδώ συνέπειες δηλαδή ε, υπάρχουν σχετικές μελέτες και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι πρόκειται περί φυσικού πάρκου που παίρνει τους πιο πολλούς κοινωτικούς πόρους για την προστασία του. Άρα, αφού ο δημόσιος Κορβανάς φροντίζει αυτό το πάρκο, από την άλλη μεριά, γιατί να δίνεται έγκριση ε, για έργα που οδηγούν στην αποθήκευση σκοέριου που φέρνει την καταστροφή αυτού του πάρκου. Θα πρέπει επομένως να υπάρξει μια πιο επικαιροποιημένη απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να καταλήξουμε στο εάν υπάρχει παράβαση όχι του δικαίου. Εντάξει, υπάρχει υπόθεση κρεμή ενώπιον των δικαστηρίων, αλλά νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να μάθουμε εάν όλα όσα γίνονται είναι σύνομα ή όχι τι γίνεται με τις οδηγίες για τα πτηνά, για το περιβάλλον, για τα ύδατα και το πιο σημαντικό είναι να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή την ερευνητική αποστολή, να πάμε οι βουλευτές στη Δονιά να, απευθυνθούμε στην Περιφερειακή Αρχή της Ανταλουσίας στις αρμόδιες αρχές τις κρατικές αρχές, τους οικολόγους, την πλατφόρμα ε, να σωθεί η Δονιάνα Νομίζω ότι πρόκειται για πρόταση όπως είπε και ο αναφέρον. Ξέρουμε ότι αυτό δεν γίνεται μέσα σε μια μέρα, αλλά θα πρέπει να κάνουμε τον προγραμματισμό μας και να κάνουμε αυτή την αποστολή τέλη του έτους ή αρχές του επομένου. Η κυρία Καμπεθών. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και τους αναφέροντες γιατί επανέφεραν αυτή την αναφορά. Νομίζω ότι ε, δεν έχει περάσει ούτε χρόνος από την τελευταία φορά. Αλλά για αυτή τη θητεία είναι η δεύτερη φορά που τα συζητούμε. Θα ήθελα να μου πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι έχει κάνει, τι έχει κάνει όλο αυτό το καιρό. Περιμένετε να αποφασίσει και να κρίνει η δικαιοσύνη. Είπαμε Κάτι πάρα πολύ απλό. Να γίνει μία μελέτη και να δοθεί απάντηση στο αν ήταν ε, νόμιμο να γίνουν οι μελέτες για το περιβάλλον αφού κόπηκε η υπόθεση στα τέσσερα χωριστά έργα. Περιμέναμε αυτό να μας πει η Επιτροπή και δεν μας το είπε. Μας επαναλαμβάνεται τα ίδια. Ότι έγινε αξιολόγηση, θετική αξιολόγηση, ε, σε δύο έργα δεν δόθηκε έγκριση, για νομικούς λόγους, ε, αλλού δόθηκε η έγκριση και ένα άλλο για διάφορους άλλους λόγους τελικά δεν έγινε τίποτα. Άρα έχουμε, τι μάθαμε, τίποτα. Τέσσερα έργα από τα οποία το ένα προχωράει και τον Ιανουάριο, το είπαμε θα πρέπει να απευθυνθούμε στις ε, διοικητικές αρχές για αυτό και ήρθε και ο ε, Επίτροπος, ο κύριος Βέλλα Ακόμα περιμένουμε την απάντηση. Στο τέλος μας είπα δεν μπορεί να κάνετε τίποτα γιατί η υπόθεση ενώπιση δικαιοσύνης έχει γίνει η καταγγελία αλλά δεν υπάρχει κάτι που να μας εμποδίζει να κάνουμε μια έκθεση σχετικά με το τι γίνεται και να υπάρξει και μια συνολική μελέτη. Τώρα έχουμε το ε, το μαρίσμο Ξιδεντάλ το έργο αυτό για το οποίο αποφάνθηκε το Πανεπιστήμιο της Σεισμολογική Μελέτη και υπάρχει και σχετική οδηγία για τι περιβαλλοντικέ επιπτώσει που επιτρέπει βάσει νέων στοιχείων να αναθεωρηθεί μια απόφαση. Άρα μπορεί και η αδειοδότηση να ανακληθεί. Άλλωστε εδώ υπάρχει και η αρχή της ε, σοφροσύνης που θα πρέπει να κυριαρχήσει. Θα πρέπει να μας ενημερώσετε για να μας ενημερώσετε εγγράφως να απευθυνθείτε και στην κυβέρνηση της χώρας. Επίσης υπάρχει και πρόταση της κυρίας Αλμπιόλ ότι θα πρέπει επιτόπου να δούμε με μια επίσκεψη τι γίνεται στην Τονιάνα γιατί είναι τεράστια η αξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτού του πάρκου. Ευχαριστώ. Πρέντα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, για την αναφορά 51, 85 του 2013, μου φαίνονται εύλογες οι ανησυχίες του αναφέροντος, όταν έχουμε ένα, μια επιχείρηση εξόριξης και μεταφοράς φυσικού αερίου πρέπει να εξασφαλίζουμε ότι δεν δημιουργούνται προβλήματα στο περιβάλλον. Από τα τέσσερα ε, έργα η Ισπανία έδωσε άδεια μόνο για ένα. Και για αυτό το ένα έχει υπάρξει προσφυγή ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων. Αυτή είναι η κατάσταση. Δηλαδή από τα τέσσερα μόνο ένα δέχθηκε, έγινε δεκτό μάλλον και, αυτό, και για αυτό πάλι υπήρξε προσφυγή στα δικαστήρια. Εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος προτείνουμε να κλείσουμε την αναφορά αυτή, γιατί η αναφορά αυτή εξετάζεται σε εθνικό επίπεδο και δεν υπάρχει τίποτα που μπορούμε να προσθέσουμε εμείς από εδώ. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος σας ευχαριστούμε. Ρόζα. Ευχαριστώ πολύ. Γνωρίζουμε ότι όλη αυτή η περιοχή εντάσσεται στο δίκτυο Natura 2000 και έχουμε την οδηγία για τους οικότοπους και για τα πτηνά και έχουμε τώρα αυτά τα τέσσερα έργα από τα οποία εγκρίθηκε από ό,τι μας λένε μόνο ένα από την περιφέρεια της Ανταλουσίας και στη συνέχεια από τις κεντρικές πανικές αρχές. Και επίσης το άλλο που ονομάζεται Μαρίσμα Οριεντάλ είπαν όχι, μία απόφαση για το Σαλαδίγιο και για το Αθναλ Καθάρ. Επίσης ε, υπερνέ η περιφέρεια της Ανταλουσίας και όχι η κυβέρνηση. Νομίζω όμω ότι δεν έχει σημασία ποιο είναι επικεφαλή τη Περιφερειακή Αρχή ή τη κυβέρνηση που είναι ο κ. Ραχώδη. Είναι θέμα τεχνικό. Και τώρα επίσης υπάρχει κάποιο είδου ε, εκκρεμωδικία, μια που είπαμε ότι το θέμα εκκρεμεί ενώπιον των δικαστηρίων. Αν όμως δεν έχει παραβιαστεί καμία οδηγία, τότε δεν υπάρχει αρμοδιότητα. Αν δεν έχουμε αρμοδιότητα, θα πρέπει να κυριαρχήσει η κοινή λογική. Να κάνουμε αποστολή εκεί. Μα αυτό, δεν το λέει αυτό η λογική. Να πάμε εάν έχουμε παραβίαση κάποιας καλά διατάξεων ή αν έχουμε αρμοδιότητα. Μα πώς να πάμε αν ε, αν ισχύουν αυτά που λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν καταλαβαίνω. Θα αποφασίσουμε όχι βάσει της λογικής, αλλά επί τη βάση της ψηφοφορίας. Πρόεδρε, ευχαριστώ, ευχαριστούμε και τους ε, αναφέροντες θα πρέπει να πούμε για άλλη μια φορά ότι είναι ένα από τα πιο σημαντικά πάρκα, από τους πιο σημαντικούς φυσικούς οικοτόπους για Ισπανία και για όλη την Ευρώπη. Και θέλει τώρα μια επιχείρηση να αποθηκεύσει εκεί όλο αυτό το φυσικό αέριο στο υπέδαφος αυτού του φυσικού χώρου. Βλέπουμε επίσης ότι διάφορες ισπανικές αρχές το 2013 ενέκριναν το έργο. Όλες μαζί. Αφού κάνανε την κατάτμιση. Μα και εγώ ερωτώ την Επιτροπή. Απευθύνθηκε στις αρχές γιατί κάνανε αυτήν την κατάτμιση και δεν έκριναν συνολικά το έργο. Να δούνε τις ε, επιπτώσεις να δουν εάν υπάρχει παράβαση του κοινοτικού δικαίου. Άρα θα πρέπει να παγώσουν τα έργα έως ότου δούμε τι συμβαίνει και να γίνει αξιολόγηση όλου μαζί του έργου και όχι του καθενός επιμέρους χωριστά. ούτε έγινε κάποια μελέτη του τρόπου διαχείρισης αυτού του έργου που να κρίνει κατά πόσον το έργο είναι ασύμβατο με το περιβάλλον. Έχει κάνει τη συμφωνία στο Παρίσι η Ευρωπαϊκή Ένωση για ε, προστασία του περιβάλλοντος, για βιώσιμες ενέργειες. Εδώ όμως κάνουμε κάτι, αυτά τα έργα αφορά ε, βρώμικη ούτως είπε ενέργεια που δεν είναι βιώσιμη ε, και επομένως κάνουμε κακό στο τόσο σημαντικό για την Ισπανία και την Ευρώπη αυτό το πάρκο κύριος του Λόγκα ε, Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε και βέβαια ευχαριστούμε και τους αναφέροντες γιατί ανέδειξαν το θέμα αυτό στην Επιτροπή μας. Η Ντονιάνα, πώς έχουμε πει τόσες φορές, δεν είναι κάτι, δεν είναι ένας χώρος, μια υπόθεση που αφορά την περιοχή της Σουέλβα ή οφρά μόνο την Ισπανία. Είναι ζήτημα ευρωπαϊκό. Ανήκει στο δίκτυο Natura 2000. Είναι ε, προστατευόμενη περιοχή από την ε, UNESCO. Αφορά τα οικοσυστήματα της περιφέρειας αλλά και όλες της Ευρώπης γιατί έχουμε πάνω από 3 εκατομμύρια πτηνά που μεταναστεύουν μέσω της Ντονιάνα προς διάφορες περιοχές Ευρώπης. Επομένως, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ακριβώς σαν ευρωπαϊκή υπόθεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που καταβάλει τόσες προσπάθειες για την προστασία της Ντονιάνα πέρσι. Εδώ στο Κοινοβούλιο είχαμε την έκθεση για την Ντονιάνα και εκεί αναφέρετο ότι έχουμε την παραβίαση του κοινοτικού δικαίου για τα, για τα ύδατα, για τους οικοτόπους, για τα πτηνά και για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Τι γίνεται τώρα με αυτές τις εγκρίσεις. Ε, εξετάστηκαν σε τέσσερις χωριστές δόσεις. Δεν έγινε μια ενοποιημένη μελέτη για τους κινδύνους από αυτά τα έργα και προγράμματα. Ο, επίσης δεν μελετήθηκε σεισμολογικά η υπόθεση γιατί είδατε τι έγινε στο, στο καστόρ της Καστελιών. Είχαμε φτάσει σε 512 ε, 512 σεισμικές δονήσεις και αυτό κόστισε σε αποζημιώσεις ένα δις. Άρα θα πρέπει και αυτό να μελετηθεί εν προκειμένου ούτε, ούτε η αρχή της ε, προλήψεως, η αρχή της σοφροσύνης ίσχυσε. Θα πρέπει να υπάρχει απόφαση για αυτή την νέα υποδομή. Είναι άγριστη. Έχουμε αυτή την αποθήκευση του φυσικού αερίου. Πρόκειται για κερδοσκοπία. Κερδοσκοπία σε σχέση με τις τιμές. Δεν είναι για να ωφελήσει κάποιον αυτή η αποθήκευση. Χουαρίστη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολύ σύντομα να σας πω ότι συμφωνώ με αυτά τα οποία ζητούν οι αναφέροντες και με αυτά που πρότειναν οι συνάδελφοι. Ακούσαμε τι έχουν να πούν και άκουσα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε θα πρέπει όντω να κυριαρχήσει η κοινή λογική. Να είμαστε επίσης προσεκτικοί και να προλάβουμε τις εξελίξεις γιατί θα είναι πολύ μεγάλη η αξία αυτού του οικότοπου, αυτού του πάρκου. Άρα θα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι τόσο εμβληματικό, τόσο ε, σημαντική αυτή η υπόθεση. Δικαιολογείται 100% το να προχωρήσει κι άλλο η Επιτροπή, να αναλύσει την υπόθεση, να μην περιμένει κανέναν. Αναμονή για πληροφορίες για το αν υπάρχει ή όχι κάποια παρανομία και όλα θα αναγίνουν πριν είναι πολύ αργά. Πρόεδρος. Σολεδάδ. Απλώς να συμπληρώσω για να αποφύγουμε κάποιες παρεξηγήσεις. Αν υπάρχουν κάποια σχέδια, κάποια έργα τα οποία θεωρείται ότι είναι αρμοδιότητα της ε, περιφέρειας, γιατί έγινε αυτή η κατάκνηση. Γιατί εξετάστηκαν χωριστά. Άρα έχει αρμοδιότητα και μπορούσε να κάνει κάτι η περιφερειακή να απευθυνθούμε και να επαναλάβουμε και προς το Υπουργείο ότι θα πρέπει να γίνει η ισορρευτική αξιολόγηση όλων μαζί των έργων. Έτσι μόνο θα τηρηθεί η νομοθεσία. Να τους ξαναπούμε ότι χρειάζεται η συνολική αξιολόγηση και να λάβουμε υπόψη για την πρόταση για την αποστολή στην Τονιάνα. No, no, no, we Δεν θα πρέπει να υπερβαίνουμε, παραβαίνουμε περισσότερες φορές. Ακούσαμε αυτό που είπατε, όλοι το άκουσαν. Αυτό που δεν καταλαβαίνω πραγματικά είναι πως όταν ακούτε ο ένας τον άλλον και επαναλαμβάνετε ο ένας τον άλλον. Γιατί δεν μπορείτε απλά να πείτε ότι προσυπογράφω αυτό που υπόθηκε για να προχωρήσουμε σε ένα νέο σημείο, με ένα καινούριο στοιχείο στο ίδιο ζήτημα, αλλά είναι λίγο τσαρλητικό να ακούμε τόσες επαναλήψεις. Είναι απίστευτο αυτό. Εξάντλησα τώρα τον κατάλογο των ομιλητών. Και ο δεύτερος αναφέρον ακόμα δεν βρίσκεται εδώ. Έρχεται, δίνω τον λόγο και πάλι στον κύριο Γκονθάλεθ για δύο λεπτά. Eh, Σύντομα. Λέτε για την κοινή λογική. Αν θέλετε τότε να εφαρμοστεί κοινή λογική, βάλτε ε, κάτω από την καθεδρική του Σαν Μάρκο ε, ένα τέτοιο χώρο αποθήκευσης. Λέμε τώρα για τη βιοπικιλότητα, για ένα μνημείο βιοπικιλότητας. Άρα ε, κατά αυτή την έννοια πρέπει να ισχύσει η κοινή λογική. Το μόνο κόμμα το οποίο θέλει αυτό το έργο είναι το Λαϊκό Κόμμα και θεώρησαν ότι είναι θετικές οι τέσσερις αξιολογήσεις. Και αυτό το έκαναν με τη ζαβολιά του να κάνουν τέσσερις χωριστές αξιολογήσεις. Υπάρχει η έκθεση που λέει ότι έχουμε ε, σεισμικό κίνδυνο. Αυτό δεν περιλήφθηκε ε, υπόψη για το μαρισμό Occidental και την έγκριση. Είπαμε για ε, ένα δις και που κάποια εταιρεία ιδιωτική σαν την, αυτή που συζητούμε τώρα έπρεπε να πληρώσει για τις δραστηριότητες μιας άλλης ιδιωτικής εταιρείας λοιπόν, που λεγόταν Καστόρ. Άρα θα πρέπει να μελετηθούν οι επενδύσεις και έχει δώσει δις αυτά που τα δις αυτά ανήκουν σε όλους τους ε, Ευρωπαίους για να προστατευτεί η Δονιάνα όχι σήμερα μόνο αλλά και στο μέλλον. Άρα θα πρέπει να πάτε, θα πρέπει να κάνετε την ερευνητική αποστολή και να δείτε από πρώτο χέρι τι λέει η Δημοτική Αρχή, τι λένε οι τρεις εμπλεκόμενες περιφέρειες της ε, Ανταλουσίας τη λέει η κοινωνία των πολιτών. Και θα δείτε πόσο οι αρχές είναι αυστηρές με τον κοσμάγι και επίοικείς με τους ισχυρούς. Και πρόκειται τώρα μην ξεχνούμε για κάποια προϊόντα τα οποία είναι κατά του περιβάλλοντος, κατά του φαινομένου του θερμοκηπίου. Έτσι θα πρέπει να γίνει η αξιολόγηση να πάτε και άμεσα να ενημερωθείτε εκεί. Δεν ενέκρινε τέσσερα. Δεν έκρινε τέσσερα Ένα, ένα, ένα μόνο ενέκρινε το, το Υπουργείο. Όχι τέσσερα, τέσσερα τότε λέει εκτό μικρόφωνου. Κοιτάξτε, δεν είναι εντελώ απαραδεκτό αυτό. Ότι επιτίθεστε σε, σε άλλα κόμματα και άλλε πολιτικέ απόψει. Εδώ πρέπει να εστιάσουμε εάν η περιοχή της Ντοράνια είναι σημαντική για σας, μην την πολιτικοποιείτε. Αυτή θα ήταν η συμβουλή μου προς εσάς και προς άλλους. Παραμείνετε στο θέμα, κρατήστε την καρδιά ζεστή αλλά το μυαλό ψυχρεμό. Είναι δυνατόν. Ο δεύτερος αναφέρον δεν έχει έρθει. Πιστεύω πως αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να προχωρήσουμε. Το επόμενο σημείο, το 21, αναφορά 1362, επειδή πρόκειται για την απαγόρευση ενοικοδόμησης σε περιοχές του δικτύου Νατούρα στη Γερμανία. Οπότε και οι Ισπανοί αναφέροντες μπορούν να δουν πως το πρόβλημα αυτό υπάρχει και σε άλλα κράτη-μέλη για να εξοικονομήσουμε λίγο χρόνο και να μην καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα πριν ακούσουμε και τον άλλο αναφέροντα. Ας προχωρήσουμε στο σημείο 21 και ξέρετε γιατί. Επειδή δεν υπάρχει κανείς αναφέρον παρόν. Εντάξει. Okay, I'm receiving εντάξει, λαμβάνω αντιφατικές πληροφορίες όλη την ώρα. Αυτό που κάνουμε τώρα είναι ότι φτάνουμε, ολοκληρώνουμε αυτήν εδώ την αναφορά που μόλις συζητήσαμε. Πριν προχωρήσουμε, άκουσα από το ΕΛΚ τι θέση να κλείσουμε την αναφορά. Άκουσα από άλλες ομάδες πως δεν θέλετε να την κλείσετε. Δεν θέλετε να την κλείσετε. Είναι προφανές αυτό. Οπότε αυτό που μπορώ να κάνω είναι να την φέρω σε ψηφοφορία. Ποιος θα ήταν υπέρ να μείνει ανοιχτή. Sí. Perdón. Hay una Συμπαθάτε με, αλλά έχει υποβληθεί μια πρόταση πρόταση για μια αποστολή, για μια επιτόπου επίσκεψη της Επιτροπής μας στην Τονιάνα. Και οι σοσιαλδημοκράτες και οι πράσινοι και οι γκουε υποστήξαμε την ε, πρόταση. Νομίζω ότι έτσι θα πρέπει να είναι η σωστή κατάληξη. Να ψηφίσουμε την πρόταση για αυτήν την αποστολή. Καθώ είστε πλήρω μέλο μέλος της Επιτροπής αυτής, θα πρέπει να ξέρετε πολύ καλά πως δεν παίρνουμε ποτέ αποφάσεις για διερμηνικέ αποστολέ σε πλήρε συνεδριάσεις, αλλά το αποφασίζουμε μεταξύ συντονιστών. Ναι, αλλά ω Επιτροπή Αναφορών θα πρέπει να αποφασίσουμε και μπορούμε, εάν η πλειοψηφία συμφωνεί γι' αυτό. Έτσι νομίζω. Συγγνώμη κύριε Σπριέδα, ζήτησε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, εγώ θα προτείνω να ακολουθήσουμε τη διαδικασία που πρότεινε, προτείνατε κυρία Πρόεδρε. Κάνατε μια πρόταση, τώρα εάν μετά ε, τίθεται μια άλλη πρόταση, εντάξει, τώρα δεν έχει νόημα να ξαναξεκινήσει η συζήτηση και να ακούσουμε ακριβώς τα ίδια επιχειρήματα. Εγώ ε, διαδικαστικά προτείνω αυτή τη στιγμή να ψηφίσουμε επί της πρότασης της Προέδρου. Soledad, I hope it's, uh, it's according to the rules. ελπίζω να είναι επί της διαδικασίας. Νομίζω δεν είναι η πρώτη φορά που η Επιτροπή μας ε, έλαβε απόφαση εδώ, στην συνεδρίαση της Επιτροπής, γιατί είναι θέμα μας, αρμοδιότητα μας. Ας πούμε για την Κύπρο. Εδώ το αποφασίσαμε και θυμάμαι και άλλες πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Γιατί ήμουν εγώ η υπεύθυνη. Εμείς οι βουλευτές πρέπει να δώσουμε μια λύση. Η πρόεδρος έκανε κάτι επί τη βάση της πλειοψηφίας των παρόντων. Νομίζω ότι η πλειοψηφία αυτό θέλει. Να ψηφίσει η Επιτροπή. Μου επιτρέπετε να πω κάτι εδώ. Ποτέ Σολεδάδ δεν πήραμε σε μια πλήρη επιτροπή με τέτοια απόφαση. Φυσικά και μπορούν να υποβληθούν προτάσει για επισκέψει στην Σουηδία, στην Ισπανία ή για διερευνητικέ αποστολέ, αλλά πάντα οι αποφάσει λαμβάνονται μεταξύ των συντονιστών. Μπορεί να προτείνεις ό,τι θέλεις, αλλά θα ήθελα να σου συστήσω πως τώρα έχουμε συνεδρίαση της Επιτροπής η οποία αναμεταδίδεται στο διαδίκτυο σε όλη την Ευρώπη. Γι' αυτό θα, θα παρακαλούσα όλοι να συμπεριφορόμαστε με τους κατάλληλους τρόπους για μια Επιτροπή. Αυτό σημαίνει πως ακολουθούμε τους κανόνες, πως βρούμε όπως σε οποιαδήποτε Επιτροπή για οποιοδήποτε θέμα και πώς προχωρούμε από αυτή τη στιγμή. Δεν πρέπει να επαναλάβω πως οι αναφορές αυτές συζητήθηκαν σε αυτή την Επιτροπή. Δύο φορές το παρελθόν. Εάν θέλετε να διατηρηθεί αναφορά ανοιχτή, πείτε το. Και στη συνέχεια προτείνετε ό,τι θέλετε στους συντονιστές εάν προτείνετε να κλείσει, όπως ο κύριος Πριέτα, τότε πείτε το, πότε θα το θέσουμε σε ψηφοφορία για να το τελειώσουμε επιτέλους. Ας προχωρήσουμε σε ψηφοφορία. Ποιος θα ήθελε να κλείσει η αναφορά. Το οποίο σημαίνει πως το ΕΛΚ είστε απομονωμένοι. Είναι αλήθεια και ποιος θα ήθελε να, διατηρηθεί, να διατηρηθούν ανοιχτές οι αναφορές SND, οι σοσιαλιστές, οι πράσινοι και η αριστερά. Είναι η πλειοψηφία. Το οποίο σημαίνει πως τώρα ας συμπεράνουμε πως η αναφορά παραμένει ανοιχτή και οι διάφορες πολιτικές ομάδες θα απευθυνθούν στους συντονιστές τους για να προτείνουν το πώς θα συνεχίσουμε. Μπορούμε να συμφωνήσουμε ως προς αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω έχουμε νέους αναφέροντες στο χώρο. Εξαιρετικά. Σολεδάδ. Eh, Κύριε Πρόεδρε, διαφωνώ. Συμφωνούμε ότι το συμπέρασμά μας θα πρέπει να είναι η πρόταση που τους συντονιστές για την ε, αποστολή και η ίδια θα είναι η πλειοψηφία και στους συντονιστές. Ήρθε εδώ ο κόσμος για να δοθεί μια λύση. Εγώ νομίζω ότι ήρθαμε εδώ και θα πρέπει, γιατί θεωρούν το θέμα σοβαρό και θα πρέπει και η απάντησή σας να είναι σοβαρή. Είναι υποχρέωσή μας να δώσουμε στον κόσμο μια απάντηση. The petition φορά αποφασίστηκε πως θα παραμείνει ανοιχτή όπως το θέλατε. Θα προχωρήσουμε αποφασίζοντας με το πως θα τη διερευνήσουμε περαιτέρω. Λάβαμε υπόψη τις προτάσεις σας οι οποίες θα τεθούν υπόψη των συντονιστών. Έτσι μπορούμε να ολοκληρώσουμε το σημείο αυτό. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο αυτή τη στιγμή για την αναφορά καθώς υπάρχουν ανοιχτές δικαστικές υποθέσεις σε εθνικά δικαστήρια. Πρέπει να περιμένουμε λίγο και τις δικαστικές αποφάσεις. Λοιπόν, τώρα ας προχωρήσουμε. Let's go. Είναι το ίδιο θέμα. Οπότε θα πρέπει να σας ενδιαφέρει. Είναι η αναφορά 907 σχετικά με την επιδείνωση των συνθηκών στο Εθνικό Πάρκο Ντονιάνα. Ο Μαντουέλ Κάντο Ρομέρα εκπροσωπεί τον αναφέροντα, τον χαιρετίζω εδώ. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας δίνω το λόγο για έως 5 λεπτά. Muchas gracias. Las marismas del Guadalquivir ocupan... Στο Γουαδαλκιβίρ είχαμε πάνω από 400.000 εκτάρια το 19ο αιώνα. Είναι ε, ρεκόρ αυτό για την Ευρώπη. Και οπότε είχαμε 35.000 που, που τώρα προστατεύονται από την Ντονιάνα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά για την τοπική πανίδα. Ε, πρόκειται για ένα από τα πιο προστατευμένα πάρκα και από την κοινωτική και από την εθνική νομοθεσία. Βρισκόμαστε επομένω τώρα σε κάποια φάση ε, κινδύνου πάρα πολύ σοβαρή. Έχουμε δύο επίση σε, δύο συνθήκες προστασίας και θεωρείται επίσης και κληρονομιά της UNESCO. Έχουμε υπόγεια ύδατα και επιφανέκα ύδατα. Και εκεί υπάρχουν πολύ σημαντικά προβλήματα. Είχαμε ένα ποτάμι από το βορρά που έχει τώρα εκτραπεί, πάει στο Γοδαλκιβίρ και από εκεί το νερό πάει εις τον ωκεανό. Πολύ λίγο νερό υπάρχει πια. Ε, οπότε έχει βουλώσει ουσιαστικά αυτό το ποτάμι τεχνητά. Και αυτό γιατί γίνονται αυτές οι φερόμενες ως παράνομες εξορίξεις. Έχουμε επίσης πάρα πολύ μεγάλη ε, ρήπανση των υδατών ε, από την εντατική γεωργία. Τώρα όσον αφορά το, τα υπόγεια ύδατα. Ε, εκεί έχουμε χρησιμοποίηση του ύδατος για κάποιου είδους παράνομες υδρεύσεις. Και η συνέπεια επίσης ήταν το ότι τώρα έχει κατέβει πάρα πολύ η στάθμη του ύδατος και είχαμε επίσης ε, ανάμιξη με αρμυρό, με θαλάσσιο νερό. Είπαν οι βεθομετρικές ότι θα πρέπει κάτι να γίνει ούτως ώστε να μπορούμε να σώσουμε αυτούς τους βιότοπους. Έχει κατέβει τώρα η στάθμη και έτσι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Επίσης, ο οικότοπος ε, ζημιώνεται πάρα πολύ από αυτό και η χλωρίδα επομένως πέραν της σπανίδας. Χάνονται τα βασικά χαρακτηριστικά του οικότοπου. και έχουν ξεραθεί επομένως τα λεγόμενα μάτια κάπου δηλαδή που έβγαινε το γλυκό νερό. Ο άνθρωπος είχε αλλάξει το περιβάλλον εδώ. Αυτό είχε πολύ αρνητικέ συνέπειες για το οικοσύστημα. Ο κίνδυνος είναι αυτονόητος. Έχουμε συγκρούσεις συμφερόντων πολιτικών και οικονομικών και έτσι δεν εφαρμόζεται ο νόμος. Το 2009, πριν από 8 χρόνια, προωθήθηκε πρώτη φορά η αναφορά αυτή και ο φορέας μας αποτελείται από επαγγελματίες που ξέρουν τι ισχύει για τα οικοσυστήματα. Είναι νομική ε, ε, και από άλλες επιστήμες. Οπότε υπάρχουν εδώ πέρα κατάφορες παραβιάσεις του δικαίου. Αδιαφορεί η κυβέρνηση και έτσι η Ντονιάνα έχει φτάσει σε οριακή κατάσταση. Αντικειμενικά, συνεχώς έχουμε βαριές παραβάσεις του δικαίου των τριών οδηγιών πλαίσιο για τους οικοτόπους, για τα νερά και για την ε, προστασία των υπογείων υδάτων από την ε, ρήπανση. Η αρμοδιότητα θεωρούμε ότι είναι αποκλειστικά κοινοτική και άρα θα πρέπει να δείξει ευαισθησία η Ένωση και το Κοινοβούλιο και απαιτήσετε την τήρηση αυτών των οδηγιών. Πριν από ένα χρόνο, το 2016, είχαμε συζητήσει και είχαμε πει ότι σύμφωνα με το 258 της Συνθήκης για την Ένωση, η Ισπανία θα πρέπει να απαντήσει στην όχληση που είχε γίνει με αιτιολογημένη επιστολή. Όμως, γι' αυτό θα πρέπει αμελητή να επισκεφθείτε την Τονιάνα θα πρέπει να είμαστε μαζί σας για να σας δείξουμε επιτόπου αυτά τα οποία ισχυριζόμαστε. Επίσης, θα πρέπει, θεωρούμε, να υποβληθεί ο φάκελος της υπόθεσης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να αποφανθεί αυτό όσο γίνεται πιο σύντομο. Ευχαριστώ πολύ. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, κ. Φερνάντες Γκόμες, είναι μαζί μας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε και ευχαριστούμε τους αναφέροντες για τα όσα είπαν. Έχουμε τώρα το, το πρόβλημα αυτό που αφορά την επιδείνωση των συνθήκων στην Τονιάνα. Αυτά έχουν διαπιστωθεί εδώ και δεκαετίες και αυτά αφορούν τις πιέσεις εις βάρος αυτού του φυσικού οικότοπου. Έχουμε μελετήσει αυτά τα οποία συμβαίνουν λόγω του ότι χρησιμοποιούνται τα ύδατα εκεί για να αποτιστούν κάποιες καλλιέργειες γιατί υπάρχει εντατική γεωργία. η γεωργία αυτή ασκείται και στις περιοχές του Natura 2000. Όπως είπε ο Αναφέρον, αναφέραμε τις καταγγελίες και καταλήξαμε στο ότι μια που δεν υπάρχουν επαρκή μέτρα για τους οικότοπους και για το Natura 2000 δεν υπάρχουν μέτρα για να υπάρξουν εγγυήσεις ούτω ώστε να πιάσουμε τους στόχους για τα ύδατα της περιοχής καταλήξαμε λέγω ότι συντρέχει περίπτωση παραβίασης της ε, νομοθεσίας για τα ύδατα και για τους οικότοπους. Άρα ξεκίνησε η διαδικασία επί παραβάση 17 Δεκάτου του 14. Η διαδικασία κατέληξε τον Απρίλιο του 16 στην Αποστολή Επιτροπής Αιτιολογημένης Γνώμης. Αναλύσαμε την ε, απάντηση της Ισπανίας για αυτή την ε, ε, αιτιολογημένη ε, απόφαση όπου είπαν ότι θα αναλάβουν τις απαραίτητες ενέργειες. Αυτό είναι η τελευταία φάση πριν το να φτάσει η υπόθεση ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Προσπαθούμε να έχουμε στη διάθεσή μας όλα τα επιστημονικά στοιχεία για να μπορέσουμε να τεκμηριώσουμε τη θέση μας εάν καταλήξουμε στο ότι υπάρχει ε, παρανομία και πριν προσφύγουμε στο δικαστήριο. Απλώς διαδικασίας επομένως έτσι έχουν τα πράγματα. Thank you very Ευχαριστώ πολύ. Γνωρίζουμε λοιπόν πως η Κομισιόν αναλαμβάνει δράση. Καλό να το ξέρουμε αυτό. Πως η Κομισιόν δεν επιτρέπει να περάσει περισσότερος χρόνος. Κύριε Πριέντα. Σας ευχαριστώ. Όσον αφορά αυτήν την αναφορά, 207, η οποία είναι από το 2009. Έχουμε φτάσει στα 8 χρόνια. Ορθώς άρχισε να κινητοποιείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη στον, τον Απρίλιο του 2016 στην Ισπανική κυβέρνηση, δηλαδή πριν από ένα χρόνο. Το ΕΛΚ ζητά να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά αυτή και ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, εργαστεί για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Ελπίζω τώρα βέβαια να μην ξαναρχίσει η συζήτηση που είχαμε πριν, γιατί τα υπόλοιπα θέματα τα συζητήσαμε και πριν. Γιατί όπως βλέπετε δεν είναι ένα θέμα που αφορά μόνο τους Ισπανούς. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Αλμπιόλ. Sí. Ε, βέβαια θα συζητήσουμε ό,τι χρειάζεται, όποτε χρειάζεται. Είτε είναι ισπανικά τα θέματα, είτε δεν είναι. Ευχαριστούμε τους αναφέροντες για το όσα μας είπαν και για το ότι ανέδειξαν το θέμα εδώ στο Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή μας και ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί σε αυτή την περίπτωση μας τα είπε ξεκάθαρα όσον αφορά τις παρανομίες, την παραβίαση του δικαίου τα πράγματα διαφορετικά σε σχέση με την προηγούμενη αναφορά. Εδώ για την Τονιάνα. Εκεί δεν μας τα είπε τόσο ξεκάθαρα όσον αφορά την αποθήκευση του φυσικού αερίου. Πάντως νομίζω ότι τώρα έχουμε μπροστά μας ακόμα μία άλλη πρόκληση. Ακόμα ένα πρόβλημα για την Τονιάνα που έχει πολλά προβλήματα. Ένα από αυτά είναι ό,τι μας εξήγησαν τώρα οι αναφέροντες. Αλλά άλλο πρόβλημα είναι αυτό που μας είπαν προηγουμένως για την αποθήκευση του φυσικού αερίου. Άρα εμείς ε, ε, ε, έτσι επιβεβαιώνουμε το ότι χρειάζεται να πάμε οι εκεί στην Τονιάνα. Και θα πρέπει με αυτή την αποστολή να μελετήσουμε όλα αυτά τα προβλήματα του Εθνικού Πάρκου. Η κυρία Καμπεθόν. Όπως είπαμε, τώρα η Επιτροπή διαπίστωσε ότι συντρέχει η αρμοδιότητά της. Αυτό αφορά τα τα εδώ, αλλά υπάρχουν περισσότερες αμφιβολίες για την αποθηκεύση του αερίου. Λέει η Επιτροπή. Εγώ νομίζω ότι τα ίδια ισχύουν και στις δύο περιπτώσεις. Θα πρέπει να εφαρμοστεί ό,τι χρειάζεται για να προστατευτεί το πάρκο. Νομίζω ότι θα πρέπει να περιοριστούν οι καλλιέργειες που είναι κοντά στην Τονιάνα. Γιατί τελικά η ζημιά προέρχεται από την ίδρυυση των καλλιεργειών εκεί. Όλα αυτά όμως θα τα δούμε άμα κάνουμε την αποστολή. Επαναλαμβάνω την πρόταση θα πρέπει να είναι το ίδιο συνεπής η Επιτροπή για όλες τις αναφορές. Ρώσο. Όταν απαντά η Επιτροπή, απαντά επί τη βάση επιχειρημάτων. Εάν σε κάποιους βουλευτές δεν αρέσκονται στα επιχειρήματα της Επιτροπής, τότε λένε ότι δεν τα λέει καλά η Επιτροπή. Τα λέει καλά όταν <coughs> αρέσουν τα επιχειρήματα. Είπε ότι δεν υπάρχει παρανομία στην μία περίπτωση και πάρει στην άλλη. Εντάξει, αφού υπάρχει εκρεμή ε, δίκη, να μην είναι ανοιχτή, είπαμε, η αναφορά. Προφανέ είναι αυτό, όπω είναι. Ε, όπως είναι επίσης λογικό το ότι δεν υπάρχουν επιχειρήματα που να στηρίζουν παρανομία. Συμφωνώ με αυτά που λέει η Επιτροπή. μια σύντομη αποσαφήνιση. Είναι η ίδια περιοχή αλλά διαφορετικά ζητήματα και η προσέγγιση σε αυτή την αναφορά είναι αμυγός επιστημονική. Είναι μια αφαιρόμενη ως παράβαση των οδηγιών για τα πτηνά, για τους οικότοπους. Δηλαδή έχουμε μια παράβαση των οδηγιών αυτών. Οπότε θα ακολουθήσουν διαδικασίες επί παραβάση. Είναι ξεκαθαρή η περίπτωση. Τώρα δίνω τον λόγο και πάλι στον κύριο Κάμπτο Ρομέρα για δύο λεπτά το πολύ. Ε, ε, Με εκπλήσει το ότι μετά από τόσα χρόνια που έγινε υποβολή, ακόμα αμφιβάλλουμε. Σας επαναλαμβάνω τι θέλουμε να έχετε τους ειδικού, τους εμπειρογνώμονες του Κλουμπ Δεντονιάνα, του, της, του μας, να έρθετε στο Εθνικό Πάρκο και εκεί θα σας εξηγήσουμε, θα σας δείξουμε ξεκάθαρα ποια είναι η κατάσταση, πώς έχει η πραγματικότητα. Γιατί νιώθουμε στο πετσί μας αυτή την, αυτή την αδράνεια, αλλά και τα όσα κουκουλώνει η κυβέρνηση, η κυβέρνηση του κράτους να έρθετε και να σας συνοδεύσουμε αποκλειστικά εμείς, το κλουμπ Ντεντονιάνα, ο φορέας μας. Thank Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι θα ήθελα να τονίσω πως εκτιμώ πάρα πολύ την επιστημονική σας προσέγγιση του ζητήματος στην αρχική σας δήλωση για την κατάσταση. Τώρα πιστεύω πως εξαντλήσαμε τη συζήτηση για το θέμα Πιστεύω πως είναι πλέον ξεκάθαρο πως θα διατηρήσουμε ανοιχτή την αναφορά και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση και επίσης καλούμε την Κομισιόν να επανελθεί με επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με το πώς προχωρούν οι διαδικασίες επί παραβάση και τι συμβαίνει. Γι' αυτό και προσδοκούμε με ανυπομονησία τη συνέχιση του διαλόγου με την Κομισιόν για το θέμα αυτό. Οπότε μπορούμε να ολοκληρώσουμε Ευχαριστώ πολύ και στον αναφέροντα κύριο Ρομέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ταξιδέψατε μέχρι εδώ και επίσης για τα ξεκάθαρα σας λόγια. Τώρα θα πρέπει να επανέλθουμε στην αναφορά 20. Ο δεύτερος αναφέροντας δεν ήρθε ποτέ. Ο, εντάξει. Ζητάτε το λόγο. Εντάξει. Ποιος είστε? Καλησπέρα μου. Αουρέλιο Κονθάλεφ. Εκπροσωπώ το Μέσα Δελαρία Δεουέλβα που είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση. Α, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ήρθατε. Καλώς ορίσατε και έχετε το λόγο. Σας περιμέναμε. Περιμέναμε να σας ακούσουμε. Έχετε το λόγο για πέντε λεπτά. Ε, πάρα πολύ σύντομα. Συγγνώμη που καθυστέρησα. Ε, υπήρχε πρόβλημα ε, στα μέσα μεταφοράς. Κατόπιν της καταγγελίας του φορέα μας το 2013 εδώ στην Επιτροπή σας σε σχέση με τις ενέργειες που γίνονται στην Τονιάνα και πάλι ήρθαμε για να σας πούμε πώς επιδεινώνονται οι συνθήκες στο Εθνικό Πάρκο γιατί υπάρχει κερδοσκοπία όσον αφορά το φυσικό αέριο στις διεθνείς αγορές είναι τρει εταιρείε που δεν έχουν καμία ευαίσθηση για το περιβάλλον. Αλλά υπάρχει και συνενοχή των αρμοδίων αρχών τη κυβέρνηση, τη κεντρική, αλλά και της, ε, των διοικητικών αρχών της Ανταλουσίας. Όλοι θέλουν να πουλήσουν σε όλη την Ευρώπη. Αυτό το έχουν ε, καταγγείλει όλοι οι οικολογικοί φορεί παντού. Και είπαμε ότι θα πρέπει εσείς να θέσετε τέρμα σε αυτή την πρακτική που βλάπτει πάρα πολύ το Εθνικό Πάρκο. Και έτσι αυτά τα έργα για την αποθήκευση ε, είναι πάρα πολύ ε, κακή ε, το κάνει η Ρεψόλ ζημιώνει το περιβάλλον και σύμφωνα με τα όσα μας είπατε επί τη βάση της απάντησης της Κομισιόν για να κλείσετε είπατε το θέμα όμως παρόλα αυτά οι αρμόδιες πανικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι η έγκριση για αυτά τα έργα δεν πρόκειται να δοθεί έως ότου δεν έχουμε την επιπλέον αξιολόγηση για τις επιπτώσεις των έργων αυτό το, παρέθεσα επιλέξει γιατί πάρα πολλά από αυτά τα έργα έγιναν χωρίς να έχουμε συνολική αξιολόγηση από πλευράς περιφέρειας και κεντρικής κυβέρνησης. Όλες, όλα αυτά τα έργα γίνονται από τρεις εταιρείες. Γκάστα του Ραλφενόσα, η Ρεψόλ και η Εναγκάς. Εσείς έχετε πλήρη τεκμηρίωση. Το 2013 σας στείλαμε όλα τα σχετικά και εμείς επαναλαμβάνουμε ότι οι αρχές είναι συνένοχοι στην επιδείνωση των συνθήκων του πάρκου. Και τώρα γίνεται επίση και επέκταση των εγκαταστάσεων των πετροχημικών τη Ουέλβα. Αρνητικές οι επιπτώσει για την Τονιάνα, ε, καταστροφικό για την λεπτή ισορροπία. Οι, οι εκεί ε, προστατεύονται από το δίκτυο το ευρωπαϊκό και ε, κανείς δεν τα προστατεύει όμως. Εδώ και δεκαετίες έχουμε στις εκβολές αυτά τα, τα εγκλήματα. Έκλεισαν κάποια ε, χωματερή, τόσο χώρο απόρριψης ε, λοιπασμάτων. Αυτά τα έκανε επιχειρηματίας που έχει μπλέξει με τη δικαιοσύνη πρόσφατα. Αυτά παραβιάζουν επίσης την οδηγία για την προστασία των υδάτων. Μέσω των διαφόρων ρευμάτων όλα αυτά τα βρώμικα ύδατα φτάνουν μέχρι το πάρκο. Ε, προέρχονται και από δηληστήρια της Ρέψα και φτάνουν μέχρι τις ακτές της Δονιάνα. Αυτά επίσης λόγω, θα γίνουν χειρότερα λόγω των έργων που γίνονται ή που θα γίνουν για το φυσικό αέριο. Επίσης, λόγω του, της φύσεως του εδάφους θα έχουμε και σεισμική δραστηριότητα όπως έγινε για το Καστόρ στην ε, Ανατολική Εκτή. Ε, και αυτό ήταν διασπάθηση του δημοσίου χρήματος για τις αποζημιώσεις, όμως εδώ τώρα τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα πλευρά σεισμολογικής. Οπότε τώρα θα έχουμε εκεί πέρα μια ορολογική βόμβα από πλευρά σεισμολογικής. Για όλα αυτά παρακαλώ κάντε αυτή την εξεταστική επιτροπή που θα πάει επί τόπου, ούτως ώστε να καταλήξουμε στα κατάλληλα και επίγοντα μέτρα για να προστατευτεί το πάρκο της Ντονιάνα που προστατεύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να αναγκάσει οι ευρωπαϊκές αρχές να παγώσουν αυτά τα έργα και να κάνουν ό,τι μπορούν για να ισχύσουν οι ευρωπαϊκές οδηγίες. Και θα πρέπει βιώσιμη ενέργεια να αναπτυχθεί και όχι να συνεχιστεί αυτό το έργο ε, για το φυσικό αέριο εκεί στα νότιο-ανατολικά της περιοχής ή το δυτικό άκρο της ε, Ευρώπης. Βέβαια εδώ παίζουν και πολιτικά παιχνίδια και μικροκομματικά συμφέροντα. Επίσης είναι πάρα πολύ προβεβλημένο το πάρκο. Έχουν γίνει ε, πάρα πολλά και ο σκοπός των κομμάτων βέβαια είναι να κερδίσουν κάποιες ψήφους. Ακούσαμε τι είπε και ο εκπρόσωπος της Ενωτικής Αριστεράς ότι στην προηγούμενη θητεία δεν έγινε τίποτα. Επί τέσσερα χρόνια από, την ε, περιφέρεια, από τις περιφερειακές αρχές. Έχουμε βαρεθεί τον οπορτουνισμό και την ε, αδράνεια των πολιτικών κομμάτων που ε, αρνούνται τις ε, ευθύνες τους. Σας ευχαριστούμε. Και ευχαριστούμε για την προσοχή που δίνεται εκεί στην ε, νότιο-δυτική γωνιά της Ευρώπης για αυτό το εθνικό πάρκο που έχει τεραστία αξία. Thank you very much. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως ήδη είχαμε μια πολύ εκτενή συζήτηση για το θέμα αυτό, πιστεύω πως πρέπει να ολοκληρώσουμε με τον ίδιο τρόπο. Θα αφήσουμε την αναφορά ανοιχτή και σας προτρέπω να στραφείτε στους συντονιστές σας. Εάν θέλετε μια διερευνητική επίσκεψη ή οποιοδήποτε άλλου είδους συνέχεια, τότε μπορούμε να το συζητήσουμε σε επίπεδο συντονιστών. Αλλά εκεί παίρνουμε σχετικές αποφάσεις. Και πάλι σχετικά με το θέμα αυτό, πολύ σύντομα, προχωρήστε. Πάρα πολύ σύντομα. Γιατί ισχύουν όλα αυτά που είπαμε προηγουμένω είπα στην ε, Κομισιόν ότι θα έπρεπε κάτι να μας πει και να απαντήσει. Αυτό ισχύει και, και εδώ. Επίσης το θέμα αυτό της κατάτμισης του έργου σε τέσσερα, να δει τι γίνεται με την ενιαία αξιολόγηση, να μας πει η Επιτροπή, δεν μας είπε. Και επίσης τι γίνεται με, τα, το σεισμολογικό πρόβλημα, ελήφθη υπόψη. Συγκεκριμένες ερωτήσεις για τους σεισμούς. Τι για να δούμε θα μπορέσει να μας ε, απαντήσει και τώρα. Τεχνικές είναι αυτές οι ερωτήσεις και συγκεκριμένες. Θα θέλατε να επανατοποθετηθείτε σχετικά έχετε να προσθέσετε κάτι σχετικά με αυτό που παρουσιάσατε για το συγκεκριμένο θέμα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα πρώτα σε σχέση με την αξιολόγηση των επιπτώσεων για αυτά τα τέσσερα έργα. Αυτό το οποίο επιτάσσει η νομοθεσία είναι το ότι όταν έχουμε περισσότερα έργα για σωρευτικά αποτελέσματα λαμβάνονται υπόψη αυτά. Όμως δεν λέει που πρέπει να γίνει μόνο μία αξιολόγηση επιπτώσεων για όλα τα έργα. Λέει ο νόμος ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη σε κάθε μελέτη τα σωρευτικά αποτελέσματα όλων των έργων και οι ισπανικές αρχές είπαν ότι για όλες αυτές τις μελέτες ελήφθησαν υπόψη τα σωρευτικά αποτελέσματα. Η Επιτροπή δεν έχει επισέτηση λεπτομέρειε γιατί μέχρι τώρα το θέμα δεν είναι κρίσιμο γιατί μόνο ένα έργο έτυχε εγκρίσιος. Άρα το θέμα αυτό δεν, δεν, δεν προσφέρει τίποτα για να το συζητήσουμε. Όσον αφορά τώρα τις σεισμολογικές μελέτες, οι αρχές της χώρας μας είπαν ότι έγινε σεισμολογική μελέτη. Και αν κάτι άλλο καινούργιο προέκυψε μετά από τις μελέτες, θα το λάβουμε υπόψη. Θα απευθυνθούμε στις αρχές της χώρας και να μας πούν πώς εκ των υστέρων θα ληφθούν υπόψη Τόσο λέει αυτή η, η μελέτη σεισμολογική και να ληφθεί υπόψη για τις συγκρίσεις. Ευχαριστώ επίσης για τις συγκεκριμένες ερωτήσεις στα μέλη της Επιτροπής. Από το ολοκληρώνουμε το σημείο 20. Ευχαριστούμε πολύ εσάς τους αναφέροντες που ήρθατε τόσο μακριά για να έρθετε εδώ στην Επιτροπή Αναφορών σήμερα πιστεύω πως πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε από αυτού με, έχει επίγοντα χαρακτήρα και με, από κοινού με τους συντονιστές θα αποφασίσουμε για τη συνέχεια και το τι θα κάνουμε αλλά είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα για το ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η παρούσα Επιτροπή είναι μια γέφυρα για τους πολίτες μεταξύ πολιτών και ευρωπαϊκών θεσμών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε και να έχετε ένα ασφαλές ταξίδι επιστροφής. Εμείς τώρα θα πρέπει να προχωρήσουμε στο επόμενο σημείο που είναι η αναφορά 1362 σχετικά με την απαγόρευση ανοικοδόμησης σε περιοχές του δικτύου Natura 2000 στη Γερμανία. Ο αναφέρον δεν βρίσκεται εδώ, αλλά η Επιτροπή όπως πάντα. Χαίρομαι λοιπόν να δώσω στον Αλεξάνδρ Τζάστ τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ο αναφέρον αναφέρεται σε δημόσιες διαθέσιμες πληροφορίες για την διαδικασία επί παραβάση δύο άρθρων της οδηγίας σχετικά με τους οικότοπους κατά της Γερμανίας ζητά να απαγορευτεί στη Γερμανία να προβεί σε κατασκευές τους τοποθεσίες αυτές μέχρι η διαδικασία επί παραβάση να κλείσει. Η Κομισιόν επιβεβαιώνει πως υπάρχει μια εκκρεμή μια διαδικασία επί παραβάση κατά της Γερμανίας σε σχέση με τον, την υποχρέωσή της να καθορίσει όλες τις τοποθεσίες υπό εθνικό δίκαιο. Το αίτημα του αναφέροντα για μια απαγόρευση ανοικοδόμησης αναφέρεται ακριβώς σε αυτές τι τοποθεσίε. Θα πρέπει να αποσαφινιστεί πως δεν απαγορεύεται η πραγματοποίηση οικονομικών δραστηριοτήτων ή κατασκευαστικών δραστηριοτήτων σε τοποθεσίε του δικτύου Natura 2000, αλλά υπό συγκεκριμένου όρους. Σύμφωνα με το άρθρο 6.3 της οδηγίας για τους οικότοπους αναφέρεται πως οποιοδήποτε σχέδιο ή έργο που μπορεί να έχει σημαντική επίπτωση σε μια τοποθεσία του δικτύου Natura θα πρέπει να υποβληθεί σε κατάλληλη αξιολόγηση των συνεπειών του και των στόχων διατήρησης. Υπό το πρίσμα της εκτίμησης, η αρμόδια εθνική αρχή θα συνενέσει σε ένα σχέδιο ή έργο μόνο αφότου εξακριβώσει πως δεν θα επηρεάσει αρνητικά την ακαιρεότητα του, της ελόγω Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 6.4 της οδηγίας, εάν παρά μια αρνητική αξιολόγηση των επιπτώσεων και αποσία εναλλακτικών λύσεων το σχέδιο ή το έργο μπορεί να πραγματοποιηθεί για επιτακτικούς λόγους και λόγω υπερέχοντος δημοσίου συμφέροντος συμπεριλαμβανομένου συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών ή οικονομικών λόγων. Το κράτος μέλος θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασπαλίσει την προστασία της συνοχής ε, της τοποθεσίας του δικτύου Natura 2000. Γι' αυτό και η Γερμανία πρέπει να εφαρμόσει τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 6.3 και 6.4 όπως και το άρθρο 6.2 το οποίο περιέχει την αρχή της μη επιδίνωσης οικοτόπων και της μη σημαντικής διαταραχής τους Συμπεραίνοντας λοιπόν η οδηγία για τους οικότοπους δεν παρέχει προβλέψεις για μια απαγόρευση ανοικοδόμησης σε περιοχές που ακόμη δεν έχουν οριστεί ως περιοχές διατήρησης σύμφωνα με τα άρθρα 6.4 και 6.3 της οδηγίας για τους οικότοπους. Τα εκάστοτε κράτη-μέλη πρέπει να εφαρμόσουν τους όρους των άφρων 6.2, 6.3 και 6.4 της οδηγίας για να, δια, για διασφαλίσουν την μη υπονόμευση της οδηγίας. Ευχαριστώ πολύ. Ανοίγει η συζήτηση. Ο κύριος Πριέντα. Ευχαριστώ πολύ. Όπως ήδη ελέγχθη, ο ανεφέρον ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαγορεύσει ουσιαστικά τις δραστηριότητες αυτέ της οικοδομικής σε μια περιοχή Natura 2000 μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν απαγορεύεται η διεξαγωγή τέτοιων οικοδομικών και οικονομικών δραστηριοτήτων ε, στην περιοχή 2000. Όσον αφορά την ε, διαδικασία, η η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας ενημέρωσε ότι έχει ξεκινήσει και είναι εξελίξει. επομένως η πρόταση του ΕΛΚΙ να κλείσει, αυτή η αναφορά. Σας ευχαριστώ. Ζητά κάποιος άλλος συνάδελφο το λόγο για το θέμα αυτό. Δεν είναι η Ντονιάνα, αλλά είναι μια άλλη ευαίσθητη, σημαντική περιοχή της Ευρώπης. Ωραία, δεν ζητά κάποιος άλλος συνάδελφος το λόγο. δεν είναι παρόν και ο αναφέρον. Θα ακολουθήσω λοιπόν την πρόταση του συναδέλφου Πρέντα. Θα ενημερώσουμε τον αναφέροντα για αυτά που διεμήφθησαν με τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα του στείλουμε μια περίληψη και ένα σημείωμα που θα εξηγεί την κατάσταση και η αναφορά κλείνει. Σας ευχαριστώ. Μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο της σημερινής διάταξης. Είναι το σημείο 22 ε, αναφορά 434 πυρηνικός σταθμός ε, Γκαρόνια στην πόλη Μπούργος. Παρευρίσκεται ο αναφέρον, αλλά και θα προσπαθήσω καλύτερα να μην... Ναι, μάλλον όχι, έχετε ζητήσει να ε, διατηρηθεί η ανωνυμία σας και βεβαίως θα τους σεβαστούμε, έχετε το λόγο για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ, πρόεδρο. Χουάν έτσι ονομάζομαι. Από μια, από μια μικρή κοινότητα προέρχομαι στο Μπούργος. Είμαι σφαντάρης. Περίπου την ίδια ηλικία έχει και αυτός ο πυρηνικός σταθμός και όλη μου τη ζωή έζησα εκεί κοντά. Σήμερα, εάν είχα ε, είχα κάτι να κάνω κάτι ήθελα να κάνω δεν θα έπαιρνα επιδότηση καμία από τη χώρα ενώ αντίθετα αυτές οι εγκαταστάσεις έχουν τύχει μεγάλων ενισχύσεων η πιο παλιά εγκατάσταση είναι δεν είναι νέα αυτή η εγκατάσταση αλλά η κυβέρνηση το μόνο το οποίο κάνει είναι να συνταξιοδοτεί αυτό το, το, το, τις γερασμένες εγκαταστάσεις. Και ξέρετε η σύνταξη δίνεται στα 67 χρόνια. Α, έτσι θα γίνει και με αυτό το εργοστάσιο. Μόνο που αυτοί ήδη έχουν περάσει σε φάση συνταξιοδότησης. Έχει κλείσει τον κύκλο της ζωής της. Από το 2012 σταμάτησαν τη λειτουργία τους. Και τώρα, και είχε αποφασιστεί επίσης από το 2013 να διαλυθεί, να γκρεμιστεί το εργοστάσιο αυτό. Είχαμε 136 συμβάντα και είπαμε ότι υπάρχουν προβλήματα στον αντιδραστήρα. Επομένως, τα 3 εκατομμύρια που ζουν εκεί κοντά κινδυνεύουν είχαμε διάφορες ρογμές εκεί και το 2004 μόλις αυτό ε, αναγνωρίστηκε. Και τελικά το είπε. Το είπαν η, η, το των χίλιων κινδύνων. Θα πρέπει να λέμε υπόψη ότι τα τρία τέταρτα των ε, αντιδραστήρων ε, πάσχουν. Δεν μπορούν να αντέξουν ένα σεισμό. Και έτσι δεν έχουν δώσει καμία λύση, μόνο προσωρινή. Αυτό όμως απαγορεύεται όσον αφορά την παραγωγή της πυρηνικής ενέργειας. Αυτές οι εγκαταστάσεις ανήκουν στην Ουκλενόρ. Είναι επικίνδυνες θα πρέπει ομιλώς να διαλυθούν άπαξ και διαπαντό, να κλείσει, να φροντίσουμε για την ασφάλεια. Τα δεδομένα δείχνουν ότι δεν έχει βοηθήσει ε, αυτή η εγκατάσταση τον εξηλεκτρισμό της χώρας. Και τώρα να ξαναλειτουργήσει αυτό το εργοστάσιο σημαίνει το να πάμε πίσω 46 χρόνια στην εποχή του ασπρόμαυρου σινεμά στην περιοχή την πιο σκοτεινή της χώρας μας. Πίσω λέει στο φραγκισμό θα πρέπει να χρησιμοποιούμε εγκαταστάσεις για καθαρή ενέργεια, ανανεώσιμη. Να έχουμε ηλιακή ενέργεια και έτσι να ε, μην ε, δίνονται άδειες και εγκρίσεις που ωφελούν μόνο τις μεγάλες εταιρείες και θα πρέπει το κράτος να σκεφτεί την ασφάλεια του περιβάλλοντος και του κόσμου. Όλα, όλα γύρω εκεί στον ε, Εύρο, στο Μπούργος, ε, προστατεύεται από το Natura 2000. Εκτός από αυτή την Χερσόνησο ε, και επομένως θα πρέπει να σκεφτούμε το πώς θα δώσουμε στην Ήπεθρο ε, κάποιες ευκαιρίες. Εμεί αυτό περιμένουμε από την Ευρώπη, αυτό θέλουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχω δύο ονόματα. Ή ο κύριος Πόπο ή ο κύριος Φλωρέα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είμαι ο κύριος Φλωρέα. Θα συνεχίσει ο κύριος Πόπο. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον κύριο Γκονθάλες, τον αναφέροντα, η Επιτροπή θα ήθελε να τονίσει πως η επιλογή μεταξύ των διάφορων ενεργειακών πηγών συμπεριλαμβανομένης της απόφασης λειτουργίας πυρηνικών σταθμών παραγωγής ενέργειας απόκειται στα κράτη-μέλη. Αν ένα κράτος μέλος όπως η Ισπανία αποφασίσει να λειτουργεί πυρηνικούς σταθμούς και αποφασίσει να παρατείνει τη λειτουργία τους πρέπει φυσικά να εκπληρώσει όλα τα κριτήρια πυρηνικής ασφάλειας σύμφωνα με την συνθήκη Ευρατών και στο δευτερογενές δίκαιο. Η ε, Κομισιόν θα ήθελε να τονίσει πως είναι ο φορέας εκμετάλλευσης, τον οποίο βαραίνει η ευθύνη, υπό την εποπτεία των εθνικών εποπτικών αρχών. η νέα τροποποιημένη οδηγία που θα μεταφερθεί έως του έως τον Αύγουστο στο Εθνικό Δίκαιο θα πρέπει να επιτευχθούν σημαντικές βελτιώσεις. Αυτό ισχύει επίσης για την περίπτωση του πυρηνικού σταθμού της Γκαρόνια και επίσης περιοδική έλεγχη ασφαλείας πρέπει να διεξάγονται μια φορά ανά δεκαετία τουλάχιστον επίσης σύμφωνα με την οδηγία περί πυρηνικής ασφάλειας. Ο Ισπανός, η Ισπανική ρυθμιστική αρχή είναι αρμόδια για την πυρηνική ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Εάν η απόφαση μακροχρόνιας λειτουργίας των εγκαταστάσεων εγκριθεί, τότε όλες οι βελτιώσεις πρέπει να υλοποιηθούν στον πυρηνικό σταθμό παραγωγής ενέργειας. Ο επενδυτής θα πρέπει να ειδοποιήσει την Κομισιόν για τα επενδυτικά έργα Εάν εκπληρωθούν τα κριτήρια, τότε είναι υποχρεωτική η ενημέρωση της Κομισιόν. Σήμερα, έως σήμερα, η Κομισιόν δεν έλαβε καμία ειδοποίηση για το σχέδιο επενδύσεων στον σταθμό της Γαρόνια. Η παρούσα ανακοίνωσή μας βασίζεται βέβαια στην συνθήκη Ευρατόμ, είναι δευτερογενές δίκαιο χωρίς να φύγεται η συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τις ε, υποχρεώσεις που ε, απορρέουν από αυτήν και το δευτερογενές δίκαιο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει τίποτα που να υποδεικνύει ότι κάτι τέτοιο θα γίνει. Εάν είναι να γίνει, πρέπει να αναφερθεί, αλλά δεν υπάρχουν κάποια στοιχεία. Έχουμε μόνο πληροφορίε από τα μέσα μαζική ενημέρωση. Τα σχέδια δεν έχουν ε, ε, ξεκινήσει ακόμα. Οπότε ανοίγω τη συζήτηση. Ο κύριος Πρετά πρώτος. Euh, ναι, ναι, εδώ. Ακόμα εδώ είμαι. Ακριβώς όπως είπατε. Δεν έγινε καμία ανακοίνωση προς την Επιτροπή. Άρα δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Και εμείς επομένως προτείνουμε να κλείσει η αναφορά. Εμείς ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Ακούστε τώρα ακολουθούν πολλά ισπανικά, ισπανοί συνάδελφοι και ο δεύτερος εκπρόσωπος της Κομισιόν πρέπει να μιλήσει ακόμα. Οπότε πιστεύω πως μπορούμε να δώσουμε το λόγο σε έναν ή δύο συναδέλφους. θελετε να μιλήσετε πρώτος, οπότε πρώτος εσείς παρακαλώ σύντομα μία μικρή αποσαφήνιση για το γεγονός ότι η Επιτροπή, η Κομισιόν απάντησε εγγράφως πολλές φορές ως προς τον πυρηνικό σταθμό. Μία τελευταία κοινοβουλευτική ερώτηση ήταν η 564 του 2017. Έχουμε μία ακόμα το 2017 την 4.1.1.7 του 2016 κτλ. κτλ η Κομισιόν απάντησε τουλάχιστον 10 φορές για τον πυρηνικό σταθμό αυτό και μάλιστα εγγράφω. Οι απαντήσεις δημοσιεύτηκαν στην ισοσελίδα μας και στο, στη σελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, εξαιρετικές πρόσθετες πληροφορίες. Για να μην μείνουμε εδώ έως τα μεσάνυχτα, παρακαλώ συνάδελφοι μην επαναλάβετε ο ένας τον άλλον και εμπνευστείτε από την τόσο ταχεία παρέμβαση του κυρίου Πρέντα σήμερα. Κυρία Βαλίνα. Ευχαριστώ. Κύριε Πρέντα. Ε, καταλαβαίνω. Θέλετε να κλείσετε όλες τις αναφορές. Αλλά... Κοιτάξτε. Λάβετε υπόψη και σεβαστείτε λίγο τις ε, ισπανικές αναφορές που για αυτές πρέπει να την χάνουν δίκη όπως όλες. Ε, δεν είναι θέμα για γέλια. Είναι επομένω η κατάσταση εδώ πέρα ανησυχητική. Γιατί έχει εξαντληθεί το όριο ζωής των εγκαταστάσεων. Σα είπα ότι έχει ομοιότητες η εγκατάσταση του, του, με τις εγκαταστάσεις της Φουκουσίμα δεν υπάρχει βιώσιμο ενεργειακό πρόγραμμα από την κυβέρνηση. Είναι υπόθεση που ε, τραβάει πολύ καιρό και το κλείσιμο των εγκαταστάσεων δεν είναι πρόβλημα για την επάρκεια την ενεργειακή στη χώρα. Πρέπει να ε, κλείσει το εργοστάσιο για να δοθούν κίνητρα για βιώσιμες πηγές ενέργειας. Να μην είναι ανοιχτή αναφορά. Να στείλουμε επιτροπή στις Ισπανικές Αρχές και να ζητήσουμε ενημέρωση όσον αφορά το πώς έχει κατάσταση ε, για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Να μην ε, προχωρήσουμε σε ενέργειες αφού ξανανοίξουν οι εγκαταστάσεις γιατί το έχουμε ξανακάνει αυτό το να επεμβαίνουμε εκ των υστέρων δεν έχει ξανανοίξει ακόμα το εργοστάσιο αλλά έτσι ανακοινώθηκε να ληφθούν μέτρα από τώρα και όχι εκ των υστέρων υποχρεούται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δίνει απαντήσεις. Ε, αν την ρωτάμε επανειλημμένα θα πρέπει πάλι κατ' επανάληψη να απαντά. Ναι, μας λέτε ότι για τις ενεργικές πηγές ε, ε, επιλαμβάνονται τα, τα κράτη. Αλλά δεν είναι αλήθεια όπως προέκυψε και, από τα, και για τα ανθρακοριχεία έχω μια πολύ μακρά, έναν πολύ μακρύ κατάλογο μιλητών και πρέπει να δώσω προτεραιότητα στα μέλη της Επιτροπής. Αλλιώς θα δυσκολευτούμε μετά. Κυρία Αλβιόλ, παρακαλώ πολύ πολύ σύντομα έτσι ώστε οι συνάδελφοι να πάρουν επίσης το λόγο. Ευχαριστώ. Δεν μιλάμε τώρα για φήμες, ούτε είναι και μαντάτα που τα μάθαμε από τις εφημερίδες η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Ασφαλείας στις 8 Φεβρουαρίου έλαβε την απόφαση αυτή για να ξανανοίξουν οι εγκαταστάσεις πυρηνικές της Γκαρόνια. Δεν πρόκειται περί φημών. Πρόκειται για αυτό το επίσημο όργανο πυρηνικής ασφαλείας. Αυτό θα είναι ιστορικό προηγούμενο. Γιατί θα εγκρίνουν παράταση ζωής πέρα από τα 40 χρόνια. θα πρέπει, λέγανε, να γίνονται κάθε 10 χρόνια ένας ε, έλεγχος της ασφάλειας. Τώρα είπα να γίνεται κάθε 14 χρόνια. Σας υπενθυμίζω όμως ότι αυτές οι εγκαταστάσεις προβλεπόταν να έχουν 25 χρόνια ζωής. Μετά η διάρκεια ζωής πήγε στα 40. Και τώρα μιλάμε για 60 χρόνια και κύκλο ζωής. Δεν χρειάζεται την ενέργεια η περιοχή είχε κλείσει προσωρινά το εργοστάσιο και δεν πρόκειψε καμία έλλειψη. Δεν είναι αναγκαία η ύπαρξη των εγκαταστάσεων. Θα πρέπει να δώσουμε περιβάλλον, στο, στο περιβάλλον προτεραιότητα και στην ασφαλειά μας. Και όχι το να κάνουν κάποιες δουλειές. Είναι αρμοδιότητα της ισπανικής κυβέρνησης, αλλά να μην ε, μας θέτει όλους εν κινδύνο. Μπορεί η Κομισιόν να πιέσει την Ισπανία να μην πάει για ε, αυτή την παράτηση ζωή στα 60 χρόνια ενό αντιδραστήρα που μοιάζει με την Φουκουσίμα. Μιλάμε για ένα περιβάλλον που προστατεύεται από το Natura 2000 να κλείσει και να κατεδαφιστεί το εργοστάσιο. Και ζητάμε από την Επιτροπή να κάνει μία μελέτη για όλες τις πυρηνικές εγκαταστάσεις στην Ευρώπη που έχουν πάνω από 40 χρόνια ζωής. Δεν είναι μόνο θέμα Ισπανίας ή της Γκαρόνια, είναι ευρωπαϊκό το πρόγραμμα. Η μελέτη για όλες τις εγκαταστάσεις. Να διαπιστωθεί σε τι κατάσταση βρίσκονται. Είπαμε δεν είναι κάτι που το μάθαμε τις εφημερίδες, είναι απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας δεν έγινε ανακοίνωση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, άρα ας απευθυνθεί η Κομισιόν στην κυβέρνηση και να ρωτήσει γιατί δεν έγινε η επίσημη ανακοίνωση για το ξανά άνοιγμα της Γκαρονιά. Η κυρία Εύβοια, Ευχαριστώ. Λαμβάνω τον λόγο για να υποστηρίξω αυτά που είπαν οι αναφέροντες Είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση. Θα πρέπει εις να μελετηθεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα όπως είπε και η συνάδελφος. Έχουμε εκεί γύρω γύρω και πολύ κοντά περιοχή του Natura 2000. Θα πρέπει κάτι να γίνει για αυτή την περιοχή. Μα ήρθε η ώρα η Ευρώπη και τα κράτη-μέλη να κάνουν κάτι συγκεκριμένο και να εγκαταλείψουν τα ορυκτά καύσιμα τις παλιές ξεπερασμένες τεχνολογίες και να προχωρήσουν προς τις ανανεώσιμες. Το 2017 είναι πολύ σοβαρό το ότι ακόμα έχουμε τέτοιες παλιές εγκαταστάσεις. Πάμε σε ουδετερότητα τεχνική. Αλλιώς με αυτό το πνεύμα οδηγόμαστε στα σκάνδαλα σαν τον Dieselgate. Θέλουμε καθαρή τεχνολογία. Επίσης είναι πρόβλημα και τι γίνεται με τα πυρηνικά απόβλητα. Να μείνει ανοιχτή αναφορά. Thank you very much. Now, Rose... Ευχαριστώ πολύ. Η Ρώσα ως πλήρως μέλος και αντιπρόεδρος της Επιτροπής θέλει να τοποθετηθεί για τον συνάδελφό της κύριο Ντιασεμέρα που δεν είναι μέλος της Επιτροπής. Παρακαλώ έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εσένα Ρώσα που μου έδωσες ε, την ευκαιρία αντί για σένα να μιλήσω. Με όλο το σεβασμό προς τους αναφέροντες θέλω να πω ανεξαρτήτως του ότι έχουμε κάποια διαφορά στην αντίληψή μας. Επίσης θέλω να, να πω ότι σέβομαι και όλες τις αντίθετες απόψεις των πολιτικών ομάδων ή κάποιες πολιτικές ομάδες, τέλος πάντων. Και ευχαριστώ και τον κύριο Πρέντα. Το πρόβλημα είναι ενεργειακό αλλά και ιδεολογικό. Πρόκειται για κρίση πολιτική αυτό είναι πρόβλημα που υπήρχε από πάντα. Δεν είναι μόνο επί του παρόντος και αναφορά μόνο την Καρόνια. Με προσοχή διάβασα την αναφορά και άκουσα τι είπε και διάβασα τι είπε και η Κομισιόν. Δεν προκύπτει παράβαση του δικαίου. Δεν δικαιολογείται ο πανικός. Απλώς υπάρχει η επισήμανση της προληπτικής δράσης. Και έχουμε τώρα το θέμα των εγκαταστάσεων και των περιβαλλοντικών συνεπειών. Έχουμε 80% ενεργειακό έλλειμμα. Δηλαδή αγοράζουμε 80% της ενέργειας που χρειαζόμαστε. 40 χρόνια είναι αλήθεια ότι έχει δουλέψει αυτό το εργοστάσιο και το κλείσανε χωρίς να είναι κάποια μελέτη και έγιναν ή θα γινόντουσαν κάποιες ε, ενέργειες για να είναι ασφαλές το εργοστάσιο. Και επίσης μας λέει ο, ο αναφέρον ότι να δούμε κατά πόσον υπάρχει παραβίαση αυτό σημαίνει ότι μπορεί να μην υπάρχει καμία παρανομία. Εάν δεν ε, προσαχθούν αποδείξεις ε, παράβασης του νόμου, ε, τότε η αναφορά μπορεί να τεθεί στο αρχείο. Μας λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι γίνεται με αυτή τη διαδικασία της ανακοίνωσης από τους ιδιοκτήτες, τους κυρίους του σχολών εγκατάστασης και ότι θα, ότι θα πρέπει να έχουν ανακοινωθεί στην Επιτροπή πώς βελτιώθηκε η ασφάλεια. Όμως η ανακοίνωση προβλέπεται μόνο εάν οι, αυτές οι αλλαγές στις εγκαταστάσεις ε, είναι συγκεκριμένου είδους και συγκεκριμένες ε, έκτασης όπως προβλέπει το κοινωτικό δίκαιο. Δεν έχει νόημα να συνεχίσουμε με αυτήν την ε, αναφορά. Άλλωστε δεν έχει νόημα κυρίως επειδή ακόμα δεν υπάρχει επίσημη απόφαση ξανά των εγκαταστάσεων. Ε, και γι' αυτό είναι αρμόδια η κυβέρνηση της χώρας. Κύριε Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω πρώτα πρώτα τον Δήμαρχο, τον ε, αναφερόμενο. Είπαμε ότι δίνεται τώρα παράταση ζωής, το αποφάσισε αυτό για λόγους πολιτικούς το, το Συμβούλιο Ασφαλείας. Όμως δεν έλαβαν υπόψη την ασφάλεια και την οικολογία. Για λόγους ασφάλειας η Γαρόνια που έκλεισε το 2013 δεν πρέπει να ξαναανοίξει. Είναι δίδυμη αδελφή αυτή η εγκατάσταση της Φουκουσίμα. Έχει πολλά προβλήματα στο σχεδιασμό των εγκαταστάσεων. Γι' αυτό και έκλεισε το 12 θέτει κινδύνο εκατομμύρια. Και θα ρηπανθεί ο ποταμός Εύρος και όλες αυτές οι περιοχές του Natura 2000. Το πρόβλημα, μάλλον η, η απόφαση του Συμβουλίου δεν ανακοινώθηκε στην Επιτροπή ε, και αυτό είναι γιατί υπάρχει πρόβλημα το σχέδιο επενδύσεων. Υπάρχει η οδηγία για την πυρηνική ασφάλεια. υπερπαράγουμε ηλεκτρισμό. Άρα να κλείσουν όλες οι σχετικές παλιές εγκαταστάσεις. Το είπε και η Μπερντρόλα ότι δεν είναι κερδοφόρα επιχείρηση η Γκαρόνια. θα πρέπει να ακολουθήσουμε τη γραμμή των καθαρών βιώσιμων ενεργειών, να απομακρυνθούμε από το πυρηνικό μοντέλο της βρώμικης ενέργειας. Να μείνει ανοιχτή η αναφορά και να διαβιβάσουμε στην κυβέρνηση της χώρας επιστολή και να πούμε ότι θέλουμε διαφάνεια να μας πούν τι γίνεται στην Καρόνια. και τι θα γίνει με όλες αυτές τις εγκαταστάσεις που αποτελούν ένα κίνδυνο τώρα γιατί έχουν ξεπεράσει τον κύκλο ζωής. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ολοκληρώνουμε τη συζήτηση οπότε θα ξαναδώσω το λόγο στον αναφέροντα, ο κύριος Ζιλουάγκα. Πολύ σύντομα παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ με όλο το σεβασμό. Ναι, σεβόμαστε όλες τις πολιτικές ε, ε, ε τάσεις αλλά να μην λέμε ψεύτικα στοιχεία. Έχουμε 147 γιγα, γιγαβάτ ως υπερπαραγωγή. Και αυτό ισχύει από το 2006 και δόθε. Ευχαριστούμε που φέρατε εδώ το θέμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μιλούμε για την τρίτη κατά σειράν πιο παλιά εγκατάσταση στην Ευρώπη. Έχω να πω για την ε, Επιτροπή ότι μας είπε ότι δεν έχει αρμοδιότητα και είναι εθνική αρμοδιότητα στο θέμα. Όμως υπάρχει μια λεπτομέρεια που το κάνει το θέμα αρμοδιότητά σας. Γιατί? Διότι τα μέτρα ασφαλείας ακόμα δεν έχουν ληφθεί. Και σύμφωνα με τις παραμέτρους που προβλέπουν οι συνθήκες και οι Euratom θα πρέπει το Συμβούλιο Ασφαλείας να διαπιστώσει ότι δεν συντρέχει κίνδυνος για να αποφασίσει. Έδωσε όμως την άδεια. Παρέτεινε τη ζωή της εγκατάστασης της Γκαρονιά. Ε, άρα τότε παραβιάζεται η νομοθεσία. Είναι επομένω θεμητό να ζητήσει κανεί από την Επιτροπή να μελετήσει το θέμα και να αναλάβει δράση. Έχουμε παράβαση της νομοθεσίας. Αλλιώς θα έχουμε τα τελεσμένα γεγονότα. Είναι γενικότερη τάση αυτή να αφήνουν τις εγκαταστάσεις να γεράσουν. Δέκα χρόνια, είκοσι χρόνια ισχύει αυτό για την καρόνια, παράταση της ζωής. Μεγάλος ο κίνδυνος για πολύ κόσμο. Και αυτό για μόνο το 1% της ηλεκτροπαραγωγής μας δεν χρειάζονται μόνο σε αυτές τις εγκαταστάσεις με τίποτα. Ευχαριστώ, Ρώσα. Όχι. Ο κύριος Κουαρίστη. Αν δώσετε τη σειρά σας στον κύριο Καμέρα, έχετε το λόγο. Απλώς, Πρόεδρε, σας επισημαίνω ότι η πηγές των πληροφοριών που επικαλέστηκε ο προηγούμενος συνάδελφος είναι τελείως διαφορετικές από τις δικές μου πηγές. Μόνο που οι δικές μου ταυτίζονται με την πραγματικότητα. Μήπως τι, δεν ξέρει ο συνάδελφος ότι δεν είμαστε νήσο συνεργειακοί. Υπάρχει ένα καλώδιο που συνδέει τη χώρα μου με την ε, Γαλλία. Δύο δις ευρώ κοστίζει και περνάει από τα Πυρηναία και, και, και περνάει από την Αραγωνία. Έχουμε 80% ενεργειακό έλλειμμα. Thank you. And now... Ευχαριστώ και τώρα πολύ σύντομα κύριε Χουαρίστη. Έχει αρμοδιότητα για τα τρόφιμα, για το περιβάλλον, για την ενέργεια. Μην το ξεχνούμε. Και ακριβώς αυτό ισχύει για την Καρόνια. Πάμε ότι είναι η τρίτη πιο παλιά εγκατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς να ξανανοίξει. Θα πρέπει να λάβει δράση η Κομισιόν. Προληπτικά. Είναι δημόσια υγεία. Είναι το τομεί αυτή που είναι πάρα πολύ Σημαντικό λόγο για να έχει αρμόδια την Κομισιόν και όχι για άλλες περιπτώσεις στρατιωτικές. Ευχαριστώ πολύ. Ας δώσουμε και πάλι το λόγο στον αναφέροντα. Υπενθυμίζω στον κύριο Βουλευτή ότι στις 6 Ιουλίου δημοσιεύτηκε το κλείσιμο. Αυτά τα πέντε χρόνια δεν έγινε τίποτα για αυτή την απόφαση για να κλείσει και να διαλυθεί το εργοστάσιο. Ακόμα περιμένουμε κάτι να γίνει με αυτές τις ανακοινώσεις. Δεν χρειάζεται για ηλεκτροπαραγωγή η γαρονιά. Εκπροσωπεί μόνο το 1% της ενεργειάς μας. Ε, καλά, αφού είμαστε τόσο ελληματικοί όπως λέτε εσείς, το 1% δεν θα μας σώσει. Thank you very much. Now. Ευχαριστώ πολύ, οπότε ας προσπαθήσουμε να συνοψίσουμε. Πιστεύω πως αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να βρούμε μία και καλή τις σωστές πληροφορίες. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε απευθύνοντα μια επιστολή στην Ισπανική κυβέρνηση και τι Ισπανικέ αρχέ, επειδή σε τελική ανάλυση πρέπει να γνωρίζουμε εάν όλα τα κριτήρια πυρηνικής ασφάλειας όπως αυτά ορίζονται στη συνθήκη Ευρατόμ πληρούνται. Και όπως τόνισε σωστά η Κομισιόν, ακόμα δεν έλαβαν καμία ειδοποίηση σχετικά με οποιοδήποτε σχέδιο επένδυσης επαναλειτουργίας του πυρηνικού σταθμού της Γαρόνιας. Οπότε πρέπει να μάθουμε, είναι ισχύει αυτό ή όχι. Γι' αυτό προτείνω να παραμείνει η αναφορά ανοιχτή και να στείλουμε μία επιστολή σε αυτούς και να τους ζητήσουμε μία ταχεία απάντηση σε μία πολύ απλή ερώτηση. Μπορεί να απαντηθεί πολύ απλά με ένα ναι ή με ένα όχι. Μπορούμε να το κάνουμε. Εντάξει. Εξαιρετικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ τον αναφέροντα που ήρθε εδώ. Εύχομαι ένα καλό ταξίδι επιστροφής στη σημείο 23 αναφορά 302 στη συνέχεια σχετικά με το χώρο υγειονομικής ταφής αποβλήτων στο Μιστερ Μπιάνκο στον Δήμο Μοντ Σάντα Αναστάσια της επαρχίας Κατάνια. Ο αναφέροντας δεν είναι εδώ, αλλά η Κομισιόν, η κυρία Άντικο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε η Πρόεδρος. Ε, θα ήθελα να ζητήσω από εκείνου που φεύγουν από την αίθουσα να μην κάνει φασαρία αν είναι δυνατόν. Ευχαριστώ. Η πρόσωπος της ε, Επιτροπής πρόκειται για ένα χώρο υγειονομικής ταφής ε, ιδιωτικό στην περιοχή Μιστερ Μπιάνκο, η ο οποίος χώρος, παρά τα μέτρα τα οποία προσπάθησαν να εφαρμόσουν οι αρχές δεν έγινε εφικτό να κλείσει, και λειτουργεί πάνω από 50 χρόνια, εξαιτίας της αντίδρασης των κατοίκων. Ο 2013 ε, ο αναφέρον υπέβαλε την προσφυγή του, την οποία ανέλησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο φάκελος έκλεισε γιατί θεωρήσαμε ότι τότε δεν μπορούσε να στοιχειοθετηθεί η καταγγελόμενη παραβίαση. Ε, δεν προσέβαλε την απόφαση αυτήν της Επιτροπής εκείνη την εποχή ο αναφέρον. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί την κατάσταση στη Σικελία και σε άλλες ε, περιοχές της Ιταλίας όσον αφορά την διαχείριση των αποβλήτων και ε, υπάρχει και μια διαδικασία επί παραβάση σε σχέση με την την κάθε έξι έτη αναθεώρηση του σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων. Έχουμε ζητήσει τα σχέδια, έχουμε μάλλον συμπεριλάβει τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων τα δημοτικά και τα περιφερειακά σε πρόγραμμα pilot και αυτή τη στιγμή αξιολογείται το, το, το σχέδιο του 2015 προσπαθώντας να δούμε κατά πόσον έχουν τηρηθεί οι υποχρεωτικές προϋποθέσεις, για παράδειγμα ο διαχωρισμός των, ε, της μορφής των αποβλήτων και επίσης ε, η υποχρέωση να κλείσουν οι χώροι υγειονομικής ταφής. Ε, το, το, το, το, αναφέρω αυτό όχι μόνο επειδή τίθεται ζήτημα τήρησης της οδηγίας πλαίσιο για την διαχείριση των αποβλήτων, αλλά επίσης για να αντιληφθούμε και ποια είναι η στάση της συγκελίας πώς σκοπεύει να διαχειριστεί τα, τα απόβλητα γενικότερα είναι τα θέματα αυτά σημαντικά, γιατί αν τα στοιχεία που τελικά λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να οδηγήσει αυτό στο μπλοκάρισμα ε, χρηματοδότησης από τα διαρθρωτικά ταμεία. Θα ήθελα να το λάβετε και αυτό υπόψη σας. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Έχουν, έχω δύο ε, ομιλητές στον καταλογό μου. Ξεκινώ με τον κύριο Πρέντα. Εμεί προτείνουμε να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά γιατί όπως ακούσαμε, είναι πιθανό να έχουν σημειωθεί παραβιάσεις του ευρωπαϊκού δικαίου περιβάλλοντος με σημαντικές επιπτώσεις για τη δημόσια υγεία ε, και να αναμείνουμε τις απαντήσεις ε, των Ιταλικών αρχών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και η κυρία Τζουφρίδα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ με αυτό που είπε η συνάδελφος να μείνει ανοιχτή η αναφορά. Με διάφορους λόγους. Πρώτα-πρώτα, γιατί προσωπικά διαπίστωσα ότι αυτός ο Χιτά είναι στην περιφερειά μου ε, Ξέρετε, εκεί είναι η γενέτειρά μου. Και οι ε, αναφέροντες ε, είπαν για το ότι δεν θέλουν και να υπάρξει άλλο χιτά και ζητούν αν είναι δυνατόν να μείνει ανοιχτή η αναφορά και να ε, συζητηθεί αρμόδιος. Το Νοέμβριο του 2013 θεωρήθηκε παραδεκτή και ξέρουμε πόση δουλειά έχει η Επιτροπή μας γιατί συζητείται η αναφορά μετά από τέσσερα χρόνια. 28 Αυγούστου του 2016. Ε, την ε, συζητήσαμε πρώτη φορά. Δηλαδή μόλις πέρσι είχαμε καινούργια στοιχεία τώρα ε, και ακριβώς ο φορέας ο οποίος ασχολείται με την περιφαλλοντική εποπτεία, η περιφερειακή δηλαδή αρχή για το περιβάλλον, αξιολόγησε τις εκπομπές από αυτήν την περιοχή και οι σχετικές τιμές των βιοαερίων είναι ανώτερες του επιτρεπωμένου. Και όσον αφορά την παρέμβαση της, ε, της Επιτροπής, είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες εγγύσεις για λειτουργία κάποιων χιτά. Εγγύσεις για προστασία περιβάλλοντος, αλλά και για την υγεία των πολιτών. Αυτό είναι και νομολογία του 10. Επίσης, δεν θα πρέπει μια χωματερή να είναι λιγότερο από 6 χιλιόμετρα από ε, κάποια πόλη, κάποια κοινότητα. Και εδώ στο Μιστρ Μπιάνκο είπαμε ότι εκεί έχουμε μια άλλη ε, εγκατάσταση χιτά και είπαμε ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι τιμές δηλαδή ακόμα και αν ε, κάποιος δεν ζει τόσο κοντά ε, ο κόσμος ανησυχεί και θέλει να προστατεύσει το περιβάλλον Τα είπαμε και σήμερα το πρωί με τον κύριο Τίμερμαντς για το ότι θα πρέπει να δείξουμε υπευθυνότητα έναντι των συμπολιτών μας. Άρα θα πρέπει να εξετάσουμε καλύτερα την αναφορά και επομένως να μην ανοιχτή. Εξαιρετικά κυρία Ήδη. Πρόεδρε ευχαριστώ. Θα πρέπει να μείνει ανοιχτή. Και εγώ το πιστεύω αυτό. η κατάσταση οδηγεί σε επιδείνωση της υγείας. Και όσο πάει πιο σοβαρή. Θα πρέπει επομένως αυτοί που ζουν εκεί κοντά να αναπνέουν ατμόσφαιρα ε, που έχει υποστεί αυτή όλη τη μόλυνση λόγω των αποβλήτων δεν έχουν υποστεί κάποια πρώτη επεξεργασία τα απόβλητα. Μεταφέρονται εκεί όσοι έχουν. Λέμε εδώ για κυκλική οικονομία, όμως δεν έχουμε εκεί πέρα κάποιο είδου ανάκτηση των πρώτων υλών κλπ. Θα πρέπει επομένω να κάνουμε το ποιοτικό άλμα και τα λόγια να γίνουν έργα. Μεγάλη ευθύνη έχουν οι τοπικές αρχές. Θα πρέπει η Επιτροπή να συνεχίσει την εποπτεία αυτών των προβλημάτων. Πρόεδρε θα πρέπει να στείλουμε επιστολή στις ε, αρχές της Σικελίας να προσέξουν το περιβάλλον και τη δημοσία υγεία. Να μας ξεκαθαρίσουν και κάποια στοιχεία, τι μέτρα έχουν ληφθεί, και τι γίνεται με την ε, ατμόσφαιρα που έχει υποστεί αυτήν όλη την μόλυνση. Επίσης θα πρέπει να τους ρωτήσουμε πότε προτίθενται να κλείσουν αυτόν τον χιτά. Να μας πούνε ακριβώς με τι χρονοδιάγραμμα θα γίνουν όλα αυτά και πότε θα καθαρίσουν την ε, περιοχή οριστικά. Ευχαριστώ πολύ και επίσης ευχαριστώ πολύ για την επικοδομητική στάση με αναφορά των μέτρων. Κύριε Κοράγια, δεν σας αναγνώρισα καν, αλλάξατε εντελώ εμφάνιση. Αυτό, αυτή είναι η βολιβιανή μου εμφάνιση. Ωραία. Εσείς ως Σουηδέζα καταλαβαίνετε ποιο είναι το πρόβλημα. Εκεί στο Μίστερ Μπιάνκο, στην Σάντα Αναστάζια, επίσης αυτές τις δύο ε, κοινότητες της περιοχής της Κατάνης. Είναι παράλογο να θεωρούμε ότι μπορεί ο κόσμος να ζήσει εκεί με αυτή την βρώμα εκεί κοντά ε, στη, στη χωματερή. Ζει κανένα στην Ολλανδία ή στη Σουηδία, στη Γερμανία, στο Βέλγιο με τέτοιου είδους συνθήκες. Αυτά είναι αδιανόητα. Ε, βέβαια να μην είναι ανοιχτή αναφορά. Να δείξουμε στους Ευρωπαίους συμπολίτε μας ότι υπάρχει η Ευρώπη και ότι υπάρχουν και θέματα για το οποίο περιβάλλον, όπως το περιβάλλον, όπως η προστασία της ε, υγείας. Είναι δυνατόν να ληφθούν μέτρα, είναι δυνατόν να ε, παρέμβουμε. Τον κορεδεύουν τον κόσμο οι περιφερειακές αρχές. στο τηρητή είπαν ότι κάτι έκαναν, είπαν θα κλείσουν την άλλη, αλλά τελικά με άλλα μέτρα και άλλα διατάγματα έμειναν και οι δύο χωματερές ανοιχτές. Είναι αδύνατο να, να αναπνεύσει κανείς εκεί. Οι συνθήκες διαβίωσης είναι απαράδεκτες. Γι' αυτό και έγινε αυτή η αναφορά. Συμφωνώ με όσο είπε η συνάδελφος Εύη, που σας εξήγησε τι μέτρα μπορεί να πάρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, όταν λέμε για διαφοροποιημένη συλλογή απορριμμάτων, ε, να έχουμε στο μυαλό μας ότι εκεί, όπως είπε και η κυρία Τζουφρίντα, και στο Μισθευγενικό έχουμε μεσιονικές συνθήκες. Πολύ πιο ψηλά τα ποσοστά. Τελικά γίνεται η διαλογή του 15%. Θα πρέπει να γίνει κάποια παρέμβαση. Και ουσιαστικά διασπαθίζονται τα χρήματα γιατί έχουμε κάποιους ιδιωτικούς χιτά. Και τώρα έχουμε ενεξελίξει δικαστικές εισαγγελικές έρευνες για αυτά. Πρόκειται για περιπτώσεις διαφθοράς και εμπλέκονται οι περιφερειακές αρχές. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να δείξει την πυγμή της η Ευρώπη να επιβάλλει στις περιφερειακές και στις εθνικές αρχές όπου χρειάζεται να κάνουν κάτι. Αυτό δεν πρέπει να κάνει για να συγκρατήσει αυτές τις ε, παραδιάσεις. Περιμένει να βρει το δίκιο του ο αναφέρον δεν είναι πολίτε δεύτερης κατηγορίας οι κάτοικοι αυτών των κοινοτήτων και αυτοί είναι Ευρωπαίοι πολίτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα μπορώ να συνοψίσω πολύ εύκολα. Έχουμε την τύχη που μία φορά έχουμε μία αναφορά χωρίς παρουσία του αναφέροντα, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει μία ομόφωνη προσέγγιση ανεξάρτητα από τις πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου θα πρότεινα να συνεχίσουμε να προχωρήσουμε ως εξή. Πρώτα απ' όλα να απευθυνθούμε στην Κομισιόν και να ζητήσουμε μια εξαντλητική απάντηση σε όλα τα αιτήματα του αναφέροντα. Με τη μορφή email θα χρειαστούμε μια πραγματική απάντηση στις ερωτήσεις αυτές. Δεύτερον, επίσης, να στείλουμε μια επιστολή στις περιφερειακές αρχές της Σικελίας, όπως είπε η κυρία Εύη, ζητώντας τους να εξηγήσουν την κατάσταση, κατά πόσο υπάρχει χρονικό περιθώριο για λιγμούς και πώς να αντιδράσουν. Και επίσης τονίζοντας πως ο σοβαρός κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία δεν είναι κάτι το οποίο ε, θα θεωρήσει ως κάτι τετριμένο το Κοινοβούλιο και πως πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε την ανθρωπινη υγεια δεν ειναι κατι το οποιο θα ζωής όλων των Ευρωπαίων πολιτών και από την σιωπή σα, καταλαβαίνω ότι συμφωνείτε να προχωρήσουμε ως εξή. Οπότε ευχαριστώ πολύ. Ας προχωρήσουμε στο επόμενο σημείο που είναι το 328 με 12 υπογραφές σχετικά με την έκθεση των εργαζομένων στη γεωργία σε γεωργικά φάρμακα. Ο αναφέρον βρίσκεται εδώ Καλώς ορίσατε κύριε Λεκαιό και επίσης κύριε Κιού. Σας δίνω το λόγο για πέντε λεπτά ο καθένας. Σας ευχαριστώ. Ε, βρίσκω... Θα, ήθελα να ζητήσω ε, από τον φίλο μου που βρίσκεται στα δεξιά μου να μιλήσει πρώτος. Λέγομαι Λογόν Κιού. Είμαι πρώην εργαζόμενος στην Ούτρια Τρισκαλιά ε, εταιρεία. επαναλαμβάνει ο μιλητής. Εργάστηκα στην εταιρεία Νοτχατρισκαλιά ε, εδώ και 20 χρόνια. Πρόκειται για μια συνεταιριστική ε, εταιρεία παραγωγή ζωοτροφών. Δηλητηράστηκα το 2009 από ένα φυτοφάρμακο το οποίο είχε απαγορευτεί από το 2007. Πρόκειται για το διχλωρβός και ε, το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί σε μεγάλες ποσότητες στην περιοχή του Πλουαζή. Το 2010 ε, έπεσα θύμα δεύτερη φορά δηλητηρίασης από ένα ε, φυτοφάρμακο το οποίο είχε άδεια αλλά παρόλα αυτά ξεπεράστηκε η μέγιστη επιτρεπτή δόση κατά 7 φορές. Μετά από αυτές τις διπλές δηλητηριάσεις ε, έχω πλέον, πάσχω πλέον από το σύνδρομο πολλαπλής χημικής αισθησίας. Αναγνωρίστηκε το γεγονός ότι ως εργατικό ατύχημα από το εργατοδικείο και υπήρξε καταδίκη σε πέντε για πέντε αδικήματα της εταιρείας. Το ζήτημα το οποίο θέτω στην Επιτροπή σας είναι να εξετάσει κατά πόσον οι γαλλικές αρχές ολιγόρησαν όσον αφορά την ε, επιτήρηση της χρήσης των φυτοφαρμάκων. Ο κύριος Λεκιό, από το 2009 η νουτρία της Τρισκαλιά και γενικότερα οι θηγατρικές του ομίλου Τρισκαλιά δημιούργησαν τεράστια προβλήματα περιβαλλοντικά με δραματικές συνέπειες για, τους, για τον πληθυσμό της περιοχής και για τους εργαζομένους της. Το 2009 για, για μια απαγορευμένη ουσία και το 2010 με αυτή την υπέρβαση της μέγιστης ε, δόσης. Σε κάθε περίπτωση, όλες αυτές τις περιπτώσεις μάλλον, οι εργαζόμενοι whistleblowers προσπάθησαν να δημοσιοποιήσουν αυτά τα σκάνδαλα με πολλά, αντιμετωπίζοντας πολλά εμπόδια. Πρόσφατα πάλι, τον Δεκέμβριο του 2016, έχουμε ένα νέο σκάνδαλο που η Τρισκαλιά αγόρασε καλαμπόκι ε, με υπερβολικές ποσότητες φωσφίνης ενός άλλου φυτοφαρμάκου και χωρίς να ενημερώσει κανέναν για αυτή την υπερβολική συγκέντρωση. Το ε, καλαμπόκι αυτό διοχετεύτηκε προ άλλε επιχειρήσει μεταποίηση που παράγουν ζωοτροφέ. Υπάρχουν τα ευρωπαϊκά κείμενα τα οποία ε, προστατεύουν του εργαζόμενου και έχουν, έχουν μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο τη Γαλλία. Ωστόσο, οι αρχέ δεν έχουν ασκήσει τα καθήκοντά του όσο έπρεπε, με αποτέλεσμα η Τρισκαλιά να μπορεί να συνεχίζει αυτέ τι δραστηριότητε με πλήρη ατιμορρησία. Θα θέλαμε λοιπόν να τεθεί το ζήτημα αυτό. Τα σκάνδαλα τη φυτοπροστασία δεν είναι μοναδικά στη Γαλλία. Είχαμε αντίστοιχα κατά τη διάρκεια του 2016 στην Ισπανία και αλλού. Ε, πρέπει λοιπόν το ζήτημα αυτό να απασχολήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τη δούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει μια έρευνα για τον τρόπο με τον οποίο οι Γαλλικέ αρχέ <coughs> έλαβαν μέτρα για την προστασία των καταναλωτών και των εργαζομένων με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο. Σα ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Πρέντα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αν έχω αντιληφθεί σωστά, δεν ήταν και πολύ ξεκάθαρο. Εάν θέλετε μπορείτε να ξαναλάβετε το λόγο να μου το διευκρινίσετε. Έχουν ήδη ληφθεί δικαστικές αποφάσεις για αυτές τις υποθέσεις. Απάντηση. Εν μέρη. Τι εννοείται εν μέρη. Ε, οι υποθέσεις είναι πολλές αφορούν πολλά, ε, πολλές περιοχές, πολλές τοποθεσίες τις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμηρος Τρισκαλιά και είχαμε μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις κάποιες προσφυγές στο εργατοδικείο, οι οποίες δικαίωσαν τους εργαζομένους αλλά. Ο κύριο Πρέντα. Ωραία. Εγώ λοιπόν αυτό που θα πρότεινα είναι να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά, ε, για να λάβουμε περισσότερη πληροφόρηση, να μάθουμε για παράδειγμα τον αριθμό των υποθέσεων, ποιε έχουν εξεταστεί από τη γαλλική δικαιοσύνη ή πιθανώς και σε άλλες χώρες, μιλήσατε για την Ισπανία πιθανώ και αλλού ε, και γι' αυτόν τον λόγο που προτείνω να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά, να λάβουμε ε, περισσότερη πληροφόρηση, να καταλάβουμε ακριβώ τι συνέβη. Ο κύριος Πρέντα, ε, θα ζητώ συγγνώμη, θα πρέπει να φύγω. Ο κύριος Γιαέρ θα έρθει να εκπροσωπήσει το ΕΛΚ στις υπόλοιπε αναφορές. Η πρόεδρος. Σας ευχαριστώ. Ε, ζητώ συγγνώμη γιατί ξέχασα να δώσω το λόγο στην εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πριν να δώσω το λόγο σε συναδέλφους βουλευτές. Αλλά από τα μάτια σας κατάλαβα ότι θέλατε να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση. Εν πάση περιπτώσει, κυρία Κορενίν, ε, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι το θέμα είναι πολύ σημαντικό. Γιατί σχετίζεται και με πολλά ευρωπαϊκά νομοθετήματα, όχι μόνο για τα φυτοφάρμακα, αλλά επίσης την οδηγία για την προστασία των εργαζομένων και την ε, έκθεση των εργαζομένων σε επικίνδυνες χημικές ουσίες. Ποιο είναι το ζήτημα εδώ. Όλοι αυτοί η ευρωπαϊκή νομοθεσία με τις διάφορες μορφές της. Και τα θέματα μάλλον που θέτουν οι αναφερόμενοι εμπίπτουν σε εθνικές αρμοδιότητες και θα εξηγήσω. Όσον αφορά τις ε, αδειοδοτήσεις για τη χρήση χημικών προϊόντων, αυτό αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών, αφού βεβαίως έχει δοθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο η έγκριση για τη χρήση της ενεργούς, ε, της ενεργού ουσίας αλλά η έγκριση για τη χρήση του φυτοφαρμάκου είναι αρμοδιότητα και ευθύνη του κράτους μέλους. Είναι επίσης αρμοδιότητα και ευθύνη του κράτους μέλους να φροντίζει για την επαρκή ετικετοθεσία έτσι ώστε οι χρήστες αυτών των προϊόντων να γνωρίζουν τι χρησιμοποιούν και ποιες μέτρα προφύλαξης θα έπρεπε να λαμβάνουν ε, η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η επιβολή κυρώσεων είναι επίσης ευθύνη των κρατών μελών με βάση την οδηγία για τα φυτοφάρμακα. Η οδηγία για τα φυτοφάρμακα έχει ως στόχο να μειωθεί ο κίνδυνος για την δημόσια υγεία και για το περιβάλλον από τη χρήση αυτών των ουσιών ε, σκαλύπτει και τη χρήση τους και την αποθήκευσή τους, αλλά επίσης και την πληροφόρηση που πρέπει να παρέχεται στους εργαζόμενους που χρησιμοποιούν τα προϊόντα αυτά. Πρόκειται για οδηγία, επομένως για άλλη μια φορά ο τρόπος εφαρμογής της εναπόκειται στα κράτη-μέλη. Από την πλευρά μας, στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχουμε ξεκινήσει έναν έλεγχο ε, όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας για την φυτοπροστασία. Ε, στη Γαλλία, ο τελευταίος έλεγχο έλεγχος διεξήχθη το 2012 και μετά το 2015 ε, όπως πολύ συχνά συμβαίνει στους ελέγχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπή, Επιτροπής, ε, καταγράφονται τα προβλήματα και ζητείτε follow-up, ζητείτε μια ε, ενέργειες να γίνουν από την εθνική κυβέρνηση που τις παρακολουθούμε εκ των υστέρων. Κάποια θέματα τα έχουν αντιμετωπίσει οι, τα έχουν αντιμετωπίσει γαλλικές αρχές, κάποια άλλα όχι και πρόκειται σύντομα η έκθεση για τη χώρα αυτή που καλύπτει τα προβλήματα που έχουν αντιμετωπιστεί και πια όχι, να δημοσιοποιηθεί. Αναφερθήκατε στην φωσφίνη. Θα ήθελα να σας αναφέρω ότι αυτή είχε απαγορευτεί από το... είχε... ήδη από το 2008. Άρα υπάρχει πρόοδος στον τομέα της απαγόρευσης ουσιών που αποδεικνύεται ότι είναι επικίνδυνες. Όσον αφορά την οδηγία για τους, τους επαγγελματικούς κινδύνους και την πιθανή έκθεση την 37 του 2004, αυτές οι οδηγίες είναι πολύ ευρείες και ζητούν και απαιτούν από τις εγκαταστάσεις, τις διάφορες επιχειρήσεις να ε, διαθέτουν μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους που χρησιμοποιούν χημικές ουσίες. Ο ορισμός είναι πολύ ευρύς, άρα μπορεί να καλύπτει και φυτοφάρμακα. Θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται οι ουσίες που ε, προκύπτουν από το διεθνές δίκαιο. Αυτό έχει γίνει και πάλι όμως αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών η εφαρμογή. Όπως είπαμε και προηγουμένως, δεν έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία να αποδεικνύουν ότι η χρήση αυτών των φυτοφαρμάκων ε, αποτέλεσε αντικείμενο εξέτασης το από τις αρμόδιες αρχές της Γαλλίας ή από το επίπεδο το δικαστικό και το οποίο θα ήταν και το πρώτο βήμα για οποιαδήποτε ενέργεια. Συμπερασματικά, πρόκειται για εθνικές αρμοδιότητες. Υπάρχει εθνική ε, συγγνώμη, ευρωπαϊκή νομοθεσία, αλλά είναι με τη μορφή οδηγιών, οι οποίε πρέπει να μεταφερθούν στο εθνικό δίκαιο και αποτελεί εθνική αρμοδιότητα η εφαρμογή του. Άρα τα ζητήματα αυτά θα πρέπει να ελεγχθούν να, σε εθνικό επίπεδο. Τώρα, όσον αφορά την, τον έλεγχο στην ε, Βρετάνη, ε, έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα ε, μια συνεργασία μάλλον μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Εθνικών Αρχών αξιολόγησης κινδύνου το οποίο καταλήγει σε ένα πολυετές σχέδιο, κάθε τόσο το αναθεωρούμε, για να είμαστε σίγουροι ότι εστιάζονται αυτοί οι έλεγχοι στους τομείς που θέτουν τους μεγαλύτερους κινδύνους. Αυτό το πολυετές σχέδιο είναι πάντοτε διαθέσιμο δημοσίως. Ε, επίσης, δεν είναι ξεκάθαρο, δεν γνωρίζουμε ακόμα ποια θα είναι τα επόμενα κράτη-μέλη τα οποία θα υποβληθούν στον έλεγχο δεν θα μπορούσαν να σα δώσω πληροφορίε σχετικά. Προεδρο. δεν θα ήταν καλή ιδέα ανάμεσα σε αυτέ τι χώρε να βρεθεί και η Γαλλία με αυτό που ακούμε. Θα ήθελα να σα ε, θέσω τα εξή ερωτήματα στα οποία νομίζω δεν απαντήσατε. Τι υποστηρικτικά στοιχεία τα οποία μα εδόθησαν τον Μάρτιο του 2017 ετέθησαν και ε, εστάλησαν μάλλον στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επιπλέον στοιχεία ε, δεν ξέρω αν απαντήσατε, αν τα έχετε αξιολογήσει αυτά τα επιπλέον στοιχεία, αυτά τα επιπλέον επιχειρήματα. Επιτροπή. Μας δώσανε περισσότερες πληροφορίες για να υποστηρίξουν τα αιτήματά τους και χρήσιμες είναι. Αλλά όλες αυτές οι πληροφορίες αφορούν τις εθνικές αρχές. Είναι και πάλι καλύπτουν αντικείμενα που αποτελούν εθνική αρμοδιότητα. Η Πρόεδρος. Άρα τις εξελογήσατε αυτές τις επιπλέον πληροφορίες, τις εξετάσατε και καταλήξατε στο συμπέρασμα ότι αυτά τα επιπλέον στοιχεία που σας εστάλησαν τον Μάρτιο του 2017 εμπίπτουν στις εθνικές αρμοδιότητες. Ωραία. Ε, τώρα η κυρία Άουκερ, απαντήσατε στο ερώτημά μου, Επιτροπή κυρία Άουκερ. Έχουμε κανόνες και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όταν παραβιάζεται το ευρωπαϊκό δίκαιο δεν μπορούμε να το αγνοούμε αυτό, να το παραγνωρίζουμε επειδή η επιχείρηση που έκανε αυτή την παραβίαση είναι μεγάλη. Ασχολούμαι με τα ζητήματα των φυτοφαρμάκων πάνω από 10 χρόνια και είπατε ότι το 2007-2008 απαγοράστηκε η ουσία. Και, και, λοιπόν, αρκεί αυτό. Δηλαδή απλώ θα έρχονται κανονισμοί για τα φυτοφάρμακα ε, και τους οποίους θα τους ψηφίζουμε και δεν θα δίνεται συνέχεια. Γιατί εδώ προσπαθούμε να απαντήσουμε σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληγεί σε τραγικό βαθμό από αυτήν την ε, απαράδεκτη συμπεριφορά ορισμένων εταιριών. Θα, θα, θα περίμενε κανείς ότι οι γαλλικές αρχές θα προσαγάγουν τους επέτειους στη δικαιοσύνη. Και να ρωτήσω και το εξή τελικά, εάν όλα αυτά είναι αντικείμενο εθνική αρμοδιότητα, γιατί κάνουμε ευρωπαϊκούς, ε, ευρωπαϊκή νομοθεσία, γιατί φτιάχνουμε ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα φάρμακα, απλώ χάνουμε το χρόνο μα, δηλαδή είναι απλώ συστάσει προ τι κυβερνήσει, παροτρύνσει. Δεν μας ενδιαφέρει να δώσουμε μια ουσιαστική απάντηση στα ζητήματα δημόσιας υγείας. Ε, επίσης, με έχουν ενημερώσει ότι οι γαλλικές αρχές αρνήθηκαν να ξεκινήσει ποινική δίωξη για, παρά την ε, ε υπερφύαλη αυτή, απαράδεκτη συμπεριφορά των υπευθύνων έναντι των εργαζομένων τους. Αν... Καλά, πρώτα απ' όλα με, με εκπλήσει το γεγονό ότι αυτή η ουσία είναι νόμιμη χρήση τη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά εντάξει. Τι λέμε στη Γαλλία, ότι αν είναι νόμιμη ουσία μπορείτε να τη χρησιμοποιείτε όπως θέλετε και δεν πειράζει να σκοτωθεί και κανένας. Εν πάση περιπτώσει, με εκπλήσει το γεγονό ότι οι γαλλικέ αρχέ δεν έχουν κάνει τίποτα για να προσεχθεί κανένα στη δικαιοσύνη για αυτή την τραγική κατάσταση. Επόμενη μιλήτρια, κυρία Χουζιέ. Σα ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και του προσ... αναφέροντε ε, και να του εκφράσω την υποστήριξή μου με τη, μετά από αυτή τη δύσκολη δοκιμασία που έχετε περάσει και σας ευχαριστούμε που μας ενημερώνετε για αυτή την κατάσταση γιατί πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο αφορά την υγεία εκατοντάδων ε, εργαζομένων και σίγουρα χιλιάδων καταναλωτών κατά βάση υπάρχει ευρωπαϊκή αρμοδιότητα η οποία αναφορά στην απαγόρευση φυτοφαρμάκων συγκεκριμένων ε, ουσιών η οποία ξεκινάει από ευρωπαϊκό επίπεδο και μετά ανατίθεται στα κράτη-μέλη. Ο έλεγχος πρέπει να γίνεται με αποτελεσματικός από τα κράτη-μέλη. Η πρόταση δική μου είναι να κρατήσουμε την αναφορά ανοιχτή για να εξετάσουμε τελικά τι αποτελεί η ευρωπαϊκή αρμοδιότητα, τι αποτελεί εθνική αρμοδιότητα και τι κάνανε οι γαλλικές αρχές ε, να δούμε πού υπήρξε το πρόβλημα. Το πρόβλημα υπήρξε στη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Ε, το πρόβλημα υπήρξε στον τρόπο που η επιχείρηση εφάρμοσε τους κανόνες ή όχι. Ε, έγιναν οι έλεγχοι. αυτέ τι πληροφορίε, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να τι έχουμε στη διάθεσή μα, ε, από ό,τι κατάλαβα επίση έχει ξεκινήσει και μια διαδικασία ε, αναγνωρίση ενάντια ε, του, του, του, του Οργανισμού κοινωνική Ασφάλισης ε, του γεγονός του εργατικού ατυχήματος. Ε, πέρα από αυτό, έχει ξεκινήσει ποινική διαδικασία. Γιατί εδώ μιλάμε για πολλές περιπτώσεις, πολλές υποθέσεις. Και θα ήθελα να μου πείτε, αν, έχετε, αν μπορείτε να το κάνετε αυτό, να μου πείτε ποιο είναι κατά τη γνώμη σα ο επιμερισμό των ευθυνών με βάση τα στοιχεία που έχετε στη διάθεσή σα. Σα ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Χαίρομαι που έχουμε παρόντες τους αναφέραντες για να μας δώσουν τη μαρτυρία τους, γιατί για τα φυτοφάρμακα γνωρίζουμε ποιε είναι οι πιθανές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και εδώ έχουμε μια συγκεκριμένη περίπτωση με έναν άνθρωπο που αρρώστησε. Και θα είδατε ότι στο εργατοδικείο, στο δικαστήριο που ασχολείται με ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης εκδικάστηκε η υπόθεση. Δηλαδή δεν υπήρξε μια ποινική δίωξη κατά του εργοδότη του, της επιχείρησης, το οποίο σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή λαμβάνει ένα επίδομα σαν να επρόκειτο για εργατικό ατύχημα, το ελάχιστο επίδομα για εργατικό ατύχημα, χωρίς να έχει γίνει μια ποινική δίωξη στον εργοδότη. Λοιπόν, εμείς εδώ είμαστε ευρωβουλευτές και ακούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είμαστε μαζί σε όλα αυτά, έτσι. Έχουμε τις οδηγίες από το 2007 λέγεται λοιπόν ότι η πρώτη ουσία, ότι ήταν, απα... ήταν απαγορευμένη. Άρα απαγορεύεται η χρήση της από μια επιχείρηση. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Μετά έχουμε και κανονισμούς. Τον κανονισμό για ε, τα υπολείμματα ε, ε, τα, τα, οποία ξεκάθαρα η μέγιστη συγκέντρωσή τους είχε ξεπεραστεί. Υπάρχει επίση ο κανονισμό 882 όσον αφορά την πρόσβαση στα επιστημονικά στοιχεία. Γιατί παρά το γεγονό ότι έγιναν επιστημονικέ έρευνε, οι εργαζόμενοι δεν είχαν πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία. Και τα λέω όλα αυτά γιατί ε, εμπιστεύομαι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά θέλω να ρωτήσω το εξή. Κάνετε ελέγχου στην περιοχή ε, Πακά και ε, Γον Αλπ. Κάτι στο πάντου καλέ. Δεν πρέπει να γίνεται και ένας, έναν έλεγχο συγκεκριμένα για την επιχείρηση Τρικαλιά. Γιατί εδώ έχουν πληγεί εκατοντάδες εργαζόμενοι. Και γιατί στέκομαι στην Τρικαλιά. Γιατί πιθανότατα πολλοί εργαζόμενοι έχουν νοσήσει πέραν από εκείνους που αυτοκτόνησαν. Επίσης είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει μια ολιγορία της γαλλικής, ε, του γαλλικού κράτους. Λυπάμαι που το λέω ως Γαλλίδα, αλλά εάν η Γαλλία είχε ε, ξεκάθαρα πει ότι η επιχείρηση η γαλλική δεν σεβάστηκε την ομοθεσία και είχε ξεκινήσει δίωξη, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Επομένως εδώ θα ήθελα να ρωτήσω επισήμως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώς κάνετε τον έλεγχο. Κάνετε έναν έλεγχο στη Βρετάνη. Τι, πώς αξιολογείτε το σεβασμό των διαφόρων ε, προβλέψεων που υπάρχουν στις οδηγίες από την πλευρά της Γαλλίας. Πιστεύετε δηλαδή ότι η Γαλλία του στηρεί τις οδηγίες και αν όχι τελικά τι γίνεται, τελικά ποιος, σε ποιον λογοδοτεί η Γαλλία εάν δεν κάνει τη δουλειά της που θα έπρεπε να κάνει. Ε, μετά. Το δικαστήριο, το εργατοδικείο, αναγνώρισε ότι επρόκειτο εδώ σε συγκεκριμένες υποθέσεις εργατικά ατυχήματα, αλλά υπάρχουν και άλλα. Και άλλε ανοιχτέ υποθέσεις. Εδώ κατά την άποψή μου αυτό που θα έπρεπε να ξεκινήσει είναι μια δικασία παραβάση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έναντι της γαλλικής κυβέρνησης για τον τρόπο με τον οποίο δεν σεβάστηκε τις ευρωπαϊκές οδηγίε Γιατί οι οδηγίε αυτέ εγκρίθηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι Γάλλοι βουλευτέ υπερψήφισαν τη σχετική νομοθεσία. Ε, αν τελικά μετά από όλη αυτή τη διαδικασία κανείς δεν επιμβαίνει, κανείς δεν παρεμβαίνει, τελικά οι εργαζόμενοι πληρώνουν. Αυτό που με ενόχλησε στην παρέμβασή σας είναι ότι σταθήκατε και επαναλάβατε πολλές φορές είναι εθνική αρμοδιότητα, είναι εθνική αρμοδιότητα. Ε, ναι, αλλά έχουμε αποδείξεις εδώ. Ακόμα και αν είναι δουλειά του νομάρχη, κάποιος πρέπει να τον αναγκάσει να ασκήσει τα καθήκοντά του εάν ολιγορεί. Επομένως δεν, δεν μου αρκεί να ακούω ότι είναι ε, εθνική αρμοδιότητα. Όταν υπάρχει μια εθνική αρμοδιότητα η οποία εκπορεύεται από ευρωπαϊκή νομοθεσία και το κράτος μέλος δεν την ε, τηρεί, κάποιος πρέπει να, να παρέμβει. Ε, εδώ μιλάμε για εργαζόμενους που τους βάλανε να ρίξουν το φυτοφάρμακο στο χωράφι χωρίς προστατευτικά μέτρα, χωρίς, χωρίς μάσκες, χωρίς τίποτα. Θα ζητήσω από τους συναδέλφους υπουργοβουλευτές να υποστηρίξουν αυτή την πρωτοβουλία και κατά την άποψή μου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία επί παραβάση. Ε, επίσης πιστεύω ότι και η Επιτροπή ε, πρέπει να πάει να κάνει έναν έλεγχο επιτόπιο γιατί η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή. Ευχαριστώ πολύ κυρία Εύη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να εκφράσω την αλληλεγγύη μου ε, προς τον αγώνα των αναφερόντων. Μαρτίου είπαμε ότι θέλουμε παραπάνω πληροφορίες. Θα πρέπει όλα τα χρήσιμα έγγραφα, όλα τα σχετικά να διαβιβαστούν. Και Σωστά σοβαρά θα πρέπει να αναλύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με μεγάλη προσοχή τα πράγματα. Έχουμε αυτές τις διαδικασίες που είναι βέβαια εθνική αρμοδιότητα γιατί αφορούν τα εθνικά δικαστήρια αλλά έχουμε εδώ και το θέμα της ε, παράβασης των ε, οδηγιών να δούμε ποιες είναι οι γαλλικές ευθύνες για αυτές τις παραβάσεις. Οπότε και τώρα πιστεύω ότι θα πρέπει η κοινότητα να σταματήσει να σταματήσει κάποιο είδους ε, γεωργία ε, κόντρα στα συμφέροντα των ε, μεγάλων ε, εταιριών εγκαταλείψης της γης. Είναι κάτι το οποίο είναι κίνδυνος για την υγεία. Και έχουμε επίσης και την ε, πρωτοβουλία αυτή για τη γλυφοσάτη. Τα είπαμε τις πρώτες και με τον κύριο Χόγκαν που μας είπε ότι χαιρέται που ε, μπορεί να προχωρήσει σε κάποια ανανέωση των σχετικών μέτρων για 10-15 χρόνια. Έχουμε όμως ε, όλες αυτές τις ε, καταγγελίες για τις τοξικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στην Γεωργία. Δεν είναι το πρόβλημα Γεωργία, θα πρέπει να είναι η λύση. Θα πρέπει να πάμε προς την ε, βιολογική Γεωργία. Οπότε επαναλαμβάνω το ότι θα πρέπει εις βάθος να εξεταστεί για να καταλάβουμε Πώς είναι δυνατόν να έχουμε περιορισμούς και, και κυρώσεις που να ισχύουν κάθε φορά που έχουμε ε, παράβαση των κανονισμών και των οδηγιών. Μαγκαρέντα, έχει μια πρόσθετη ερώτηση. Επειδή δεν το κατάλαβα πριν, όταν διαβάζουμε στην απάντησή σας προς εμάς, παραθέτω, όσον αφορά το προϊόν αυτό η Επιτροπή αποφάσισε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να μην το εγκρίνει το 2007. Τα κράτη-μέλη μπορούν να δώσουν μια περίοδο χάριτος η οποία πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομη και να λύγει το αργότερο την έκτη Σεπτεμβρίου 2008. Τι σημαίνει αυτή η πρόταση, αν είναι εθνική αρμοδιότητα, να αποφασίσουν. Και πιστεύω πως μπορώ να γίνω επίσης λίγο πιο απότομη από τη συνάδελφός μου. Όπως ακούσαμε ότι ο αναφέρον δηλητηριάστηκε το 2009, προφανώς οι γαλλικές αρχές δεν έκαναν τίποτα. Ποια είναι η απάντησή σας σε αυτό. Μπορώ να έχω το λόγο. Σημαίνει πως η ουσία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά από την μεταβατική περίοδο αυτή. Αυτό σημαίνει. Εάν συμβεί κάτι, κάτι με άλλον τρόπο σε ένα κράτος μέλος, αυτό είναι αρμοδιότητα αυτού του κράτους μέλους. Το πρώτο βήμα θα ήταν να προσφύγει κανείς, να απευθυνθεί μάλλον στο κράτος μέλος έτσι ώστε αυτό να πάρει τα κατάλληλα μέτρα. Αυτό μπορεί να γίνει σε εθνικό επίπεδο. Από τους ανθρώπους που έχουν συνείδηση αυτού. Παραδείγματο χάρη. Αφετέρου, η Κομισιόν κάνει ελέγχου. Πρέπει να πω πως δεν συμμετέχω άμεσα σε αυτό. Και οι έλεγχοι αυτοί γίνονται ανατακτά χρονικά διαστήματα, καλύπτουν διαφορετικά κράτη-μέλη, τα προγράμματα αποφασίζονται με πολυετή βάση και η επόμενη σειρά ελέγχων συζητείται όσον αφορά ποια κράτη, σε ποια κράτη-μέλη, σε ποιες περιφέρειες, ποια στοιχεία θα πρέπει να ελεγχθούν. Αυτό είναι ακόμα ανοιχτό και συζητείται και φυσικά και θα ενημερώσουμε για τη σημερινή συνεδρίαση. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε θέση να σας ενημερώσω, επειδή το ζήτημα είναι πολύ πιο περίπλοκο η λήψη των αποφάσεων, δηλαδή ποιοι θα είναι οι έλεγχοι. Αλλά μπορώ να προσθέσω πως η έλεγχοι αυτή για τη χρήση φυτοφαρμάκων και τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων δεν σχετίζονται άμεσα με τις οδηγίες για την προστασία των εργαζομένων. οι οποίες καταρτίζονται από την Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης. Φυσικά και υπάρχουν κάποιες σχέσεις. Εκεί θα μπορούσαμε να έχουμε μια αλληλεπικάλυψη όσον αφορά τη χρήση φυτοφαρμάκων. Όσον αφορά την ερώτηση τι σημαίνει έχουμε ενωσιακό δίκαιο και εθνικό δίκαιο. Ίσως θα έπρεπε να το ξεκαθαρίσω λίγο περισσότερο. Έχουμε την έγκριση των δραστικών ουσιών σε ενωσιακό επίπεδο. Εάν μια ουσία εγκριθεί αυτό σημαίνει πως ένα προϊόν φυτοπροστασίας που περιέχει την ουσία αυτή μπορεί να εγκριθεί σε ένα κράτος μέλος ένα κράτος μέλος δεν μπορεί να εγκρίνει προϊόντα φυτοπροστασίας με δραστικές ουσίες που δεν έχουν εγκριθεί. Συμφωνώ ως προς αυτό και είναι καταρχάς εθνική αρμοδιότητα. Εμείς ελέγχουμε. Αλλά η διαδικασία χορήγησης έγκρισης πρέπει να γίνει σύμφωνα με ενιαίέ αρχέ τη Ευρωπαϊκή Ένωσης. Δηλαδή το κάθε κράτος μέλος δεν μπορεί να εγκρίνει προϊόντα όπως θέλει ή σύμφωνα με τις προτεραιότητε του, αλλά πρέπει να ακολουθήσει το ενωσιακό δίκαιο βάσει ενιαίων αρχών, ενιαίων κινδύνων, έτσι ώστε να ληφθεί η απόφαση κατά πόσον θα μπορεί να εγκριθεί η χρήση ενός συγκεκριμένου μέσου προστασίας. Πρόεδρος. Πιστεύω πως εξαντλήσαμε το θέμα, πρέπει να ολοκληρώσουμε. Υπάρχουν διάφορα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Θα δώσω πρώτα τον λόγο πίσω στον αναφέροντα. Παρασύρθηκα κι εγώ. Ορίστε, έχετε το λόγο για δύο επιπλέον λεπτά. Σας ευχαριστώ. Σήμερα αυτό που θα θέλαμε να κάνουμε είναι να κρούσουμε τον κόδωνα του κινδύνου, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν θύματα. Είναι τραγική κατάσταση, πρόκειται για μια καταστροφή για το περιβάλλον, για τη δημόσια υγεία. Αλλά πέρα από αυτό υπάρχει και το συμβάν του Δεκεμβρίου του 2016. Στείλαμε νέα στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που πραγματικά ήταν η τελευταία σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Το οποίο πραγματικά μας οδηγεί να είμαστε εξοργισμένοι με τον τρόπο με τον οποίο δηλαδή να, να ρωτιόμαστε τελικά ποιο είναι αυτό που εμποδίζει τι ε, γαλλικέ αρχέ να κάνουν τη δουλειά του. Η επιχείρηση Τρισκαλιά είναι από τις πιο επικίνδυνες. σε μια ουσία η οποία έχει καταγγελθεί, είναι γνωστές οι, οι κίνδυνοι που εγκυμονεί στείλαμε, στείλαν οι ίδιοι εργαζόμενοι επιστημονικές αναλύσεις, έγιναν επιστημονικές αναλύσεις από την επιχείρηση και αρνήθηκαν οι υπεύθυνοι της επιχείρησης να μοιραστούν με τους εκπροσώπους μας στο συνδικαλιστικό μας φορέα τα στοιχεία αυτά τα επιστημονικά. Ε, μόνο για να πάρετε μια εικόνα για το τι, συνολική, για το τι ε, συμβαίνει σε αυτή την εταιρεία. Σας ευχαριστώ, η Πρόεδρος. Νομίζω μπορούμε ομόφωνα να συμφωνήσουμε ότι η αναφορά θα παραμείνει ανοιχτή και θα λάβουμε τα εξή βήματα. Πρώτον, θα στείλουμε επιστολή γραπτός στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητώντας να διεξαχθεί όσο το δυνατόν συντομότερα ένας έλεγχος στη Γαλλία. Ε, βεβαίως δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το πράξει, αλλά μπορούμε να το ε, προτείνουμε να κάνουμε μια σύσταση. Δεύτερον, θα στείλουμε μια επιστολή στις Εθνικές Αρχές της Γαλλίας υπογραμμίζοντας αυτό που μόλις είπε ο, προσφε... Ε, αναφέρον, ότι χρειαζόμαστε επιστημονικά στοιχεία, ότι χρειαζόμαστε πλήρη πληροφόρηση ε, για να γνωρίζουμε τι έχει κάνει η Γαλλία, πού βρίσκεται η κατάσταση στη Γαλλία αυτή τη στιγμή. Και το, η επιστολή επίσης πολύ προσεκτικά θα επισημαίνει ότι το δικαίωμα στην υγεία και η προστασία της δημόσιας υγείας είναι, αφαρμόζεται ομοιόμορφα σε ολόκληρη την Ευρώπη και γι' αυτό το λόγο μπορούμε να εκφράσουμε για την κατάπληξή μας για το γεγονό ότι ακόμα δεν έχουν ε, εναρμονιστεί με την οδηγία Μάργαρετ εγώ ακόμα δεν έχω καταλάβει ακόμα πώς είναι δυνατόν, είναι νόμιμο να χρησιμοποιείται ένα προϊόν το οποίο συμπεριλαμβάνει μια μία εγκεκριμένη ουσία. Γιατί ξαφνικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας είπε ότι είναι, είναι εθνική αρμοδιότητα η χρήση μιας μη εγκεκριμένης ουσίας. Ε, Βεβαίω πρώτα πρέπει να απευθυνθούμε στη Γαλλία, αλλά αν η Γαλλία αρνηθεί, δεν πρέπει, δεν οφείλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει δράση κατά της Γαλλίας από τη στιγμή που είναι παράνομη η χρήση μιας μια εγκεκριμένη ουσίας. Η πρόεδρος βεβαίως θα μπορούσαμε να συζητήσουμε τις νομικτικές πτυχές του, του, του θέματος. Νομίζω όμως χρειαζόμαστε το εξή. επιπλέον στοιχείο στη συζήτηση ότι εδώ δεν μιλούμε για κανονισμούς, μιλάμε για οδηγίες. Ε, και παραμένει το, το πρόβλημα βέβαια, αλλά ε, το 2008 δόθηκε μια περίοδος χάριτος, μάλλον έληξε η περίοδος χάριτος και ξεκάθαρα κάποιες επιχειρήσεις συνέχισαν να χρησιμοποιούν φυτοφάρμακα με αυτή την ουσία αρκετό καιρό μετά την λήξη της περίοδου χάριτος, άρα κάτι σοβαρό έχει συμβεί εδώ και πρέπει να το ελέγξουμε. Μπορούμε να κλείσουμε τη συζήτησή μας εδώ. Σας ευχαριστώ. Ε, θα ήθελα να απευθυνθώ και σε εσά. Ε, ήρθατε από όχι και τόσο μακριά ε, σε σχέση με του άλλου πολίτε που ήρθαν από την Ισπανία που μόλι έφυγαν. Σα δεν ήταν και τόσο μεγάλο το ταξίδι σας. Παρόλα αυτά, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την επιμονή σα για το γεγονό ότι υποβάλλατε αυτή την αναφορά, ότι ήρθατε εδώ, ότι είχατε αυτή την ανταλλαγή απόψεων, αυτή την παρουσίαση σε εμά. Σα ευχαριστώ πολύ και καλό ταξίδι επιστροφή. Ας περάσουμε στο σημείο 25, πάλι γαλλικό θέμα. Ποιότητα του αέρα δεν είναι μόνο τα φυταφάρμακα είναι και η ποιότητα του αέρα στην ε, Γαλλία. Είναι η αναφορά 2467 του 2014, δεν είναι παρόν ο αναφέρον. Είναι, είναι παρούσα όμως εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, Μάρτα Μουνιός Κουέστα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να στα πω στα ισπανικά. Να σας ενημερώσω για την απόφαση της 30ης Μαρτίου του 2016. Ναι, η ατμόσφαιρα είναι πρόβλημα. Και γι' αυτό και έχουμε ένα σώμα νομοθεσίας. Έχουμε τις σχετικέ οδηγίες και την ενισχυμένη οδηγία για τις οριακές τιμέ. Το Γεμβρίου του 2016 όμως, παρόλα αυτά υπάρχουν λόγια ανησυχία οι σχετικές πολιτικές μας οδήγησαν σε κάποια πρόοδο όσον αφορά τις εκπομπές. Και έχει βγούμε βελτιώσεις και στην Γαλλία συγκεκριμένα. Έχουμε την έκθεση του 16. Δείχνει ότι η Γαλλία από το 1990 μέχρι το 2014 είχε κατά το μείωση του διοξιδίου του αζότου και των άλλων εκπομπών. Και επίσης έχουμε τις εκπομπές του αμμονίου που έχουν αυξηθεί όμως. Και όπως τα λέει και στην αναφορά και είναι κάτι της υπηρεσίας περιβάλλοντος του 16 είχαμε κακή ποιότητα και αύξηση πρόωρων θανάτων στη Γαλλία. Συγκεκριμένα λέμε ότι 45.120 πρόωρες θάνατοι αποδίδονται σε αυτά τα νανοσωματίδια και 1.800 και τέτοιοι θάνατοι αφορούν το όζον και περίπου 8.000 και κάτι θάνατοι πρόωροι οφείλονται στο διοξίδιο του αζότου. Και όλα αυτά γιατί είχαμε υπέρβαση των ηριακών τιμών. Το 2005 είχαμε την ετησία έκθεση και αναφέρθηκαν σε 15 ζώνες ε, υπέρβαση και σε 6 τα νοσοματίδια και επίσης σε μία κατηγορία είχαμε υπέρβαση των τιμών νανοσωματιδίου και για το διοξίδιο του αζότου επίσης έξι κατηγορίες και στο Παρίσι που αφορά αυτή η έκθεση και αυτά όσον αφορά τα νανοσωματίδια επίσης είχαμε υπέρβαση στο Παρίσι. Εμείς παρακολουθούμε από κοντά την εξέλιξη της υπέρβασης των τιμών στην Γαλλία και σε όλα τα κράτη-μέλη που αναφέρουν υπερβάσεις. και πάντοτε αντιδρούμε με την διαδικασία επί παραβάση. Έχουμε επίσης τη διαδικασία της αιτιολογημένης γνώμης για τα διοξίδια του αζότου. Ο κύριος Γιάρ εκτός μικροφώνου. Α, θέλετε να σας τα λέω πιο σιγά. Θέλετε να συνεχίσω ή, ή να πάω παρακάτω. Α, παρακάτω, παρακάτω. Να με συγχωρούν οι διερμηνείς, γιατί μιλάω τόσο γρήγορα. Όπως έλεγα, το Φεβρουάριο του 2017 προχώρησε σε αιτιολογημένη γνώμη η Επιτροπή όσον αφορά το διοξίδιο του αζότου και τις υπερβάσεις σε 19 σημεία και στο Παρίσι και στη Μασαλία μεταξύ αυτών. Επίσης τον Απρίλιο του 2015 υπήρξαν οι υπερβάσεις, η εκθέση για την υπέρβαση των νοσοματιδίων σε διάφορες ε, περιοχές και στο Παρίσι και στη Μασαλία. Τώρα τα κράτη-μέλη διαλέγουν τα μέτρα, αλλά μπορούμε να υποδείξουμε ορισμένα, ας πούμε, κάποια μέτρα για τις εκπομπές από την ενέργεια και από την καύση ορυκτών ε, καυσίμων σε γεωργία, σε μεταφορές, μείωση της κυκλοφορίας, αλλαγή των ε, καυσίμων και επίσης ε, να υπάρξουν άλλοι κανόνες οδήγησης. Αυτό αφορά και την ε, οδηγία για τις ουριακές τιμές εκπομπών σε επίπεδο εθνικό. Η επιλογή των μέτρων πάντως, η τελική επιλογή είναι αρμοδιότητα εθνική ε, βέβαια και δεν ήταν αρκετά τα όσα έγιναν ούτω ώστε να συμμορφωθούν τα κράτη για τις οριακές τιμές της οδηγίας. Και έτσι έγινε, σε αυτό κατέληξε η αξιολόγηση της έκθεσης της Γαλλίας των ημερομηνιών που είπαμε. Οπότε επί τη βάση αυτών των ετησίων εκθέσεων λάβουμε υπόψη και τις ε, απαντήσεις για να δούμε αν θα προχωρήσουμε προς ε, διαδικασία επί παραβάση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανοίγει η συζήτηση για τους συναδέλφους. Πέτερ, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σε αδρές γραμμές διαφαίνεται, αν και η αναφορά προέρχεται από τη Γαλλία, πως υπάρχουν επίσης προβλήματα σε άλλα κρατημέλη. Το γνωρίζω και από τη δική μου χώρα, πως και εκεί υπάρχουν προβλήματα, πως ξεσπάνε μεγάλες αντιμαχίες για σε σχέση με τους δημοτικούς φορείς οι οποίοι πολλές φορές αισθάνονται μόνοι τους επειδή χρειάζονται όπως υποστηρίζουν επιστημονική συνοδεία για το πως με βιώσιμο και εντατικό τρόπο μπορεί να βελτιωθεί η ποιότητα του αέρα. Γι' αυτό και χαίρομαι που έχουμε μία παρακολούθηση σύμφωνα με την Κομισιόν ότι το πρόβλημα είναι γνωστό στις Βρυξέλλες και αν κατάλαβα σωστά Υπάρχει μια διαδικασία επί παραβάση. Αυτό σημαίνει πως η αναφορά πρέπει να παραμείνει ανοιχτή και θα περιμένουμε τι θα συμβεί. Επειδή στην αρμόδια Επιτροπή Περιβάλλοντος θα περιμένουν κάτι τέτοιο, ίσως πρέπει να το να παραπέμψουμε την αναφορά εκεί, επειδή πρόκειται για μια οδηγία που προέρχεται από τον περιβαλλοντικό τομέα. Ε, προσωπικά δεν ξέρω ακριβώς τι η προσωπική μου απόψη είναι ότι δεν ξέρω τι πήγε στραβά. Υπάρχουν κάποιες τιμές και όταν μιλάω με φορείς λήψης αποστάσεων στο δημοτικό επίπεδο μου λένε ότι έχουμε κάνει ό,τι, ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε. Έχουμε εξαρτήσει τις δυνατότητές μας, η γεωγραφική μας θέση είναι αυτή που είναι. Ή θα απαγορέσουμε την κυκλοφορία ή δεν ξέρουμε πια τι να κάνουμε. Δηλαδή χρειάζεται οπωσδήποτε μια επιστημονική συνοδεία με την έννοια της επιστημονικής βοήθειας έτσι ώστε να επιτύχουμε τον κοινό μας στόχο, δηλαδή τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα. Αυτό που είναι τόσο εύκολο εκ των, ε, εκ των έξω, αγαπητοί οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, κάντε κάτι. Αυτό είναι αρκετά περίπλοκο και αν ενημερωθείτε στον γερμανόφωνο χώρο Ιδίω ο Δήμο τη Στουτγκάρδη, στη Βάδη Βιερτενβέργη, έχει τεράστιο πρόβλημα και ο Δήμαρχο είναι πράσινο. Δηλαδή το ζήτημα δεν είναι πολιτικό. Ο αέρα δεν είναι πολιτικό. Δηλαδή κάποιε φορέ δεν είναι τόσο εύκολο να λυθεί το πρόβλημα. Γι' αυτό και πιστεύω πω η αναφορά πρέπει να παραμείνει ανοιχτή και να μεταβιβαστεί στην Επιτροπή Περιβάλλοντο, η οποία και, θα... και η Επιτροπή θα συνεχίσει να ασχολείται με το ζήτημα όπω και στα προηγούμενα χρόνια. pour indiquer, je pense qu'effectivement, on a, de ce que je... Ναι, ακόμη βρίσκονται εξελίξει σχετικέ έρευνε. Είναι γενικευμένο το πρόβλημα, άρα να μην η αναφορά. Okay, then let's do that. Let's keep the petition open. Οπότε ας το κάνουμε έτσι, ας κρατήσουμε την αναφορά ανοιχτή. Η κυρία Εύη, επίσης παρακαλώ. Sì, eh, solo και εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να μείνει ανοιχτή η αναφορά. Και γιατί σήμερα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος μιλήσαμε για τη στρατηγική της Ένωσης για την βιώσιμη κινητικότητα. Να ξανατονίσουμε ότι είναι σαν θάλαμη αερίων η πόλη μας. και είχαμε αυτό το σκάνδαλο με την, ε, με το, με την κατηγορία των αυτοκινήτων, το, το ευρώ τις διάφορες κατηγορίες τέλος πάντων για τις εκπομπές των αυτοκινήτων και είχαμε το σκάνδαλο Volkswagen οπότε και θα πρέπει να αναλυφθεί πραγματική δράση το συντομότερο ε, όχι να σταυρώνουν τα χέρια μου συνήθως γιατί η ποιότητα της ατμόσφαιρας είναι δικαίωμα και θα πρέπει να προσεχθεί ως δικαίωμα. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσει η Επιτροπή τις ελεγκτικές αρμοδιότητες ακριβώς όπως προβλέπεται και στα πλαίσια της διαδικασίας επί παραβάση. Αλλά θα πρέπει η Επιτροπή να εξετάζει και τα αυτοκίνητα. Τώρα είπαμε θα πρέπει να αναθεωρηθεί η οδηγία για την πιστοποίηση να κάνουμε κάτι απτό και να μπει φρένο σε αυτές όλες τις απάτες που είσαι οι καταναλωτές και είναι τόσο για την υγεία. Ευχαριστώ πολύ και τώρα ολοκληρώνουμε. Σήμερα πω πώς θα κρατήσουμε, όπω είπαν και όλοι, πώς θα κρατήσουμε την αναφορά ανοιχτή και θα γράψουμε επίσης ή μάλλον θα περιμένουμε λιγάκι και όταν υπάρξει νέα κυβέρνηση στη Γαλλία θα του στείλουμε μία επιστολή ιδίω στον νέο Υπουργό Περιβάλλοντος της Γαλλίας έτσι ώστε να του επιστήσουμε την προσοχή στο ζήτημα αυτό και θα του ή της αναφέρουμε ε, πως παρακολουθούμε στενά το τι συμβαίνει. Εάν Υπάρχουν δύο διαδικασίες επί παραβάση κατά της Γαλλίας. Αυτό αποτελεί ένδειξη του ότι δεν μπορούμε απλά να αφήσουμε το ζήτημα, αλλά πως πρέπει να ασχοληθούμε με περισσότερο βάθος. Και επίσης πρέπει να το στείλουμε στην Επιτροπή Ένβη. Φυσικά και δεν μπορούμε να τους διατάξουμε να παράξουν οτιδήποτε, αλλά μπορούμε να επιστήσουμε την προσοχή τους στο θέμα και ίσως έχουμε μια γνωμοδότηση από αυτούς. Εντάξει, μπορούμε να το κάνουμε έτσι εξαιρετικά. Από τη Γαλλία τώρα στη Φινλανδία αναφορά 192 σχετικά με την πρόσβαση σε έγγραφα και περιβαλλοντικές πληροφορίες. Δεν βρίσκεται κανείς αναφέρον εδώ, αλλά ο εκπρόσωπος της Επιτροπή, Ευρωπαϊκής Επιτροπής βρίσκεται εδώ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αυτή η αναφόρα αφορά την πρακτική του Εθνικού Δασοκομικού Κέντρου της Φιλανδίας που δεν παρέχει τα δεδομένα, τις πληροφορίες που χρειάζονται σχετικά με την βιοποικιλότητα σε δάση. Η Κομισιόν άρχισε τη δική της έρευνα επί του ζητήματος και το 2015 κίνησε μια διαδικασία επί παραβάση. Η Κομισιόν εξέδωσε την πρώτη προειδοποιητική επιστολή το 2015 και στη συνέχεια το 2016 τη δεύτερη. Η Φιλανδία θεωρεί πως το σύστημα διαχείρισης δασοκομικών δεδομένων είναι παρόμοιο με αυτό των προσωπικών δεδομένων. Και αυτό για τον λόγο ότι τα δεδομένα αυτά μπορούν να βρεθούν εύκολα στο, στο σύστημα διαχείρισης δασοκομικών δεδομένων. Καθώς στο σύστημα αυτό είναι μεταξύ άλλων καταχωρημένοι και οι ιδιοκτήτες των δασών. Γι' αυτό και η Φιλανδία θεωρεί πως τα δεδομένα αυτού του Μητρώου μπορούν να αποκαλυφθούν μόνο από συγκεκριμένε συνθήκες. Η Κομισιόν θεωρεί πως οι φιλανδικές αρχές μεταχειρίζονται όλα, τα δεδομένα στο Μητρώο αυτό ως προσωπικά δεδομένα και πως αυτή η ερμηνεία δεν είναι συμβατή με το ενωσιακό δίκαιο καθώς κάποιες από τις πληροφορίες αυτές πληρούν τις προϋποθέσεις για να θεωρηθούν περιβαλλοντικές πληροφορίες οι οποίες σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο θα πρέπει να κατασταθούν προσβάσιμες. Όσον αφορά την δεύτερη προειδοποίηση στη διαδικασία επί παραβάση, η Φιλανδία σηματοδότησε την διαθεσιμότητά της να τροποποιήσει την ε, νομοθεσία της έχει υπάρξει ένα αντίστοιχο νομοσχέδιο και στις 24 Μαρτίου φέτος έχει υπάρξει μια νομοθετική πρόταση. Η Κομισιόν επιτρέπει τη διαφάνεια με την οποία το αρμόδιο Φιλανδικό Υπουργείο επεξεργάζεται την υπόθεση αυτή και βρισκόμαστε σε επαφή με τις φιλανδικές αρχές για να διασφαλίσουμε τη σωστή εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. για μία φορά υπάρχει μία Σουηδέζα εκπρόσωπος της, της Κομισιόν και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Η συζήτηση έχει ανοίξει για τους συναδέλφους. Η κυρία Στανόκα πρώτα, όχι, δεν ζητήσατε το λόγο. Εντάξει, εντάξει. Πέτερ. Ίσως συμφωνήσουμε πολύ γρήγορα. ποτέ δεν μου δόθηκε αφορμή για να αφισβητήσω τα λεγόμενα της Κομισιόν. Μπορούμε να κλείσουμε την αναφορά επίσης επειδή έχουν εκπληρωθεί τα πάντα. Υπάρχει ένας υπόλοιπος κίνδυνος, αλλά θα μας ενημερώσει η Κομισιόν. Στην περίπτωση που στην τελική ευθεία η Φιλανδία στρίψε αριστερά ή δεξιά, αλλά από ό,τι κατάλαβα τώρα, υπήρξαν εντόνες συζητήσεις με τη Φιλανδία και η Φιλανδία δήλωσε η Κομισιόν μάλλον δήλωσε ότι αυτό δεν είναι στο πνεύμα της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και η Φιλανδία επέστρεψε στο έδαφος του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Η αισιόδοξη δηλαδή θα λέγαμε ας, το ας την κλείσουμε, η απεσιόδοξη ίσως είναι λίγο δύσπιστη να θέλουν να το δουν πρώτα γραμμένο με γραπτή μορφή, οπότε για να δούμε τι λένε οι συνάδελφοι. Εγώ θα έλεγα την κλείνουμε. Είμαι ε, ο αισιόδοξο της Επιτροπής δεν αμφισβητώ τις ε, αρχές. Πρόεδρος, αλλά κανείς άλλος δεν ζήτησε το λόγο. Μία φορά η κυρία Εύη. Τότε εγώ είμαι απεσιόδοξη και προτιμώ να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά μέχρι να δω σε γραπτή μορφή αποτελέσματα. Και για μία φορά συμφωνούμε πλήρως με τον Πέτριάκ επειδή πιστεύω πως πρέπει να κρατήσουμε ανοιχτή την αναφορά, αλλά όχι για πολύ καιρό, επειδή ακούσαμε από την Κομισιόν πως θέλουν να περιμένουν οι φιλανδικές αρχές να τροποποιήσουν το εθνικό δίκαιο με δέοντα τρόπο Γι' αυτό και θα έλεγα να συγκρατήσουμε ανοιχτή και να έχουμε μια συνέχεια για το ζήτημα. Θα έλεγα να στείλουμε μια επιστολή στη φιλανδική κυβέρνηση, λέγοντά του πώ συνεχίζουμε να έχουμε ένα μάτι ανοιχτό ω προ αυτό που συμβαίνει στη Φιλανδία. Εντάξει, τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπότε τελειώνουμε με τα σημεία της υπηρεσίας διάταξης. Σας εύχομαι καλό βράδυ.